is appalling. We do have uh, uh, we do have uh, an un it works now? Oh, well, here we go. Also, dann kann ich in meiner Muttersprache. Μάλιστα, λοιπόν, να συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα, λέει ο πρόεδρο. Η σημερινή ανεργία που πλήττει την Ευρώπη έχει φτάσει υψή ε, απαράδεκτα 10% σε κάποιες χώρες, πολύ υψηλότερα σε κάποιες άλλες. Έχουμε μεγάλα προβλήματα με τους ε, νέους 20% έχει φτάσει το ποσοστό της ενεργείας στους νέους και 40% σε κάποιες χώρες όπως η Ισπανία και αυτό φυσικά περιορίζει και ασκεί πίεση περιττέρω στους ήδη ε, περιορισμένους προϋπολογισμούς γιατί μειώνονται και οι σφορές. τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη έχουν συνδράμει στην ε, αναχέτηση του κοινωνικού αντίκτυπου της ανεργίας αυτής. Παρ' όλα αυτά όμως ε, τίθεται απέτηση να προβούμε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις των κοινωνικών συστημάτων στην Ένωση τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε μακροπρόθεσμα την αγορά εργασίας για να διασφαλίσουμε ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα παραμείνει ισχυρή και θα αυξηθεί και θα πρέπει κυρίως, και γι' αυτό χαίρομαι που έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Μόντι, θα πρέπει να ενισχύσουμε εκ νέου την εσωτερική αγορά. Εθνικοί προστατευτισμοί και οι σε ε, οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και μπορεί να υπόσχονται βράχει πρόθεσμα επιτυχία, αλλά σίγουρα δεν αποτελούν μακροπρόθεσμα τη σωστή λύση. Βρισκόμαστε σε μια φάση δημογραφικής αλλαγής ταχύτατης και θα πρέπει να αναζητήσουμε νέους, ε, νέες οδούς ε, και σε ό,τι αφορά την ε, υγειονομική περίθαλψη και ίσως να μας φανούν χρήσιμες λύσεις όπως η ηλεκτρονική υγεία και το γεγονός ότι μάλλον το, η εστίαση σε κοινωνικά θέματα δεν αποτελεί μόνο ευρωπαϊκό θέμα και ο πρόεδρος Ομπάμα χτες ε, υπογράμμισε το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα της Προεδρίας τους και δήλωσε ότι θέλει να αφιερώσει στον κλάδο αυτό 30 επιπλέον δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που μαστίζουν το τομέα. Έχετε την ημερήσια διάταξη για σήμερα. Δεν ε, θέλω, δεν έλαβα μάλλον καμία αίτηση για τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. Τώρα λοιπόν ε, που δουλεύει και η τυρμηνία, να σας πω ότι έχουμε τυρμηνία σε 17 γλώσσες. Δεν έχω άλλες ανακοινώσεις να κάνω, γι' αυτό λοιπόν να περάσω κατευθείαν στο πρώτο σημείο στην διάταξη. Όπως σας είπα, έχουμε σήμερα τη μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας τον Μάριο Μόντι ως πρώτο ομιλητή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος ε, του Έγκυρου Πανεπιστημίου Μποκόνη στο Μιλάνο. Ήταν πρώην ε, Ευρωπαίος ε, Επίτροπος Ανταγωνισμού και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Ήταν ισχυρός ε, υπέρμαχος της ενιαίας αγοράς ως την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην παγκοσμιοποίηση και γι' αυτό λοιπόν επαναδιορίστηκε από τον πρόεδρο Ομπάμα για να διεξάγει μία μελέτη αναφορικά με την ενιαία αγορά και την εξάρτηση του δυναμικού της. Έχετε το λόγο κύριε Μόντι. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Introductory. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τολμηρή απόφαση που έλαβε να συστήσει αυτή την Επιτροπή. Και να σας συγχαρώ και προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, και την εισηγήτρια, την κυρία Περβάους Περές, αλλά και τα μέλη της Επιτροπής για κάτι που με εντυπωσίασε πολύ από τα μέχρι τώρα πεπραγμένα της Επιτροπής. Διαπιστώνω ότι τα προγράμματά σας είναι πραγματικά βαρισίμαντα και μπορεί η Επιτροπή σας να μην έχει νομοθετικές αρμοδιότητες, αλλά σίγουρα έχει ισχυρές διανοητικές και πολιτικές ε, εξουσίες και θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξέλθει από την κρίση, ίσως την τραβήξει και από την κρίση. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης αυτής. Τα έξι μέλη των δύο θεματικών ενωτήτων που θα υποδεχθούμε εντό ολίγου είναι διακεκριμένες προσωπικότητες ε, με επιστημονική και πήρα και πραγματογνωμοσύνη και εμπειρογνωμοσύνη για τα θέματα αυτά και η δική μου πρόσκληση οφείλεται στο ότι όπως είπατε και εσείς έχω και εγώ κάποια πήρα σε θέματα ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα η εσωτερική αγορά ήταν από την πρώτη μέρα που ήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 1995 για την πρώτη ακρόαση που ήρθα εδώ Είχα πει και είχα αισθανθεί ότι το θέμα της ε, ολοκλήρωσης αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ε, κοινωνίας, της ε, κοινωνικής οικονομίας. Αυτό το είχα αισθανθεί από την αρχή και εξακολουθεί να αποτελεί ακράδα την πεποίθησή μου. Εγώ λοιπόν θα ασχοληθώ με την κρίση και ιδιαίτερα με, την, τον κοινωνικό της αντίκτυπο σε σχέση με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της αγοράς. Με δύο λόγια, η άποψή μου είναι ότι η κρίση δημιούργησε όχι μόνο τεράστια προβλήματα στην οικονομία και στην κοινωνία, για να μην αναφέρουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και σοβαρότατα προβλήματα στην διαδικασία της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Ταυτόχρονα όμως, η κρίση αυτή, αν την χωνέψουμε κατά κάποιο τρόπο διανοητικά και εκεί θα μας βοηθήσετε εσείς για να γίνει αυτή η πέψη, μπορεί να δημιουργήσει και ευκαιρίες. Η κρίση μπορεί να δημιουργήσει τις ευκαιρίες και τις προϋποθέσεις για μία νέα όθηση με πιο ισορροπημένο όμως και αποδεκτό τρόπο της διαδικασίας ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Αν λοιπόν καταφέρουμε να εξέλθουμε αισιόδοξα και δραστήρια από την κρίση, μπορεί να καταστήσουμε την ολοκλήρωση πιο συμβατή με τους ρητούς και πια στόχους της συνθήκης της Λισαβόνας, προκειμένου να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μία ε, οικονομία, κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλή ανταγωνιστικότητα. Και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ λίγο. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας επιτάσσει να γίνουμε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς άκρος ανταγωνιστική. Θα ήθελα όμως να θέσω μια ομοία ερώτηση. Δύναται η Ευρώπη να γίνει μια τέτοια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Ας είμαστε ειλικρινείς. Εγώ προσωπικά ομολογώ ότι δεν γνωρίζω, δεν ξέρω αν κάποιος από εσά γνωρίζει πώς είναι δυνατόν να χειριστούμε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς σε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί παρόλο που δεν είναι εύκολο, γνωρίζουμε πώς μπορούμε να χειριστούμε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς ε, ε, στη, σε εθνικό επίπεδο και η μεταπολεμική Γερμανία, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, υπόδειγμα μάλλον, για το πώς κανείς μπορεί να έχει μια άκρος ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς σε εθνικό επίπεδο. Εκεί περιορίζονται μέχρι στιγμής οι εμπειρίες μας. Μπορούμε όμως να πούμε σοβαρά και έγκυρα ότι το ίδιο μπορούμε να το μεταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή μια ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς. Δηλαδή μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συμπεριλάβουμε υψηλές δόσεις κοινωνικής οικονομίας στην αγορά. Μήπως αυτές οι δόσεις κοινωνικής οικονομίας παρεμποδίσουν την ολοκλήρωση της αγοράς και αναχαιτήσουν την πορεία της προς την ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι από διανοητική άποψη και από θεωρητική άποψη το ερώτημα αυτό είναι βαρισίμαντο. Εγώ αντιλαμβάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα δοχείο που σταδιακά και χάρη σε όλα τα κράτη-μέλη της δέχεται εισρωές <laughs> που με την άδεια σκύρια θα έλεγα ότι προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία. Γιατί καταφέραμε να χτίσουμε την Ευρώπη με την ε, ανεκτήμητη βοήθεια αρχικά της Γερμανίας, ε, της Γαλλίας, της Ιταλίας και τους άλλους ιδρυτές, αλλά χρησιμοποίησαμε τη γερμανική εμπειρία για να χτίσουμε αυτή την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Και συμπεριλάβαμε και το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας ήδη από τη συνθήκη της Ρώμης του 1957. Για να μην πούμε για τη συνθήκη Χάλιβα και Άνθρακα. Και μετά είχαμε το τμήμα της κοινωνικής οικονομίας αγοράς που περιλάμβανε και τη δημοσιονομική ισορροπία, το χαμηλό πληθωρισμό, μία ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα και μετά περάσαμε στην Ευρώπη όπως διαμορφώθηκε από τη συνθήκη του Μάστριχ. Τώρα η συνθήκη της Λισαβόνας είναι ακόμη πιο φιλόδοξη. Λέει ότι θέλουμε την πλήρη κοινωνική οικονομία της αγοράς. Πώς όμως συνδυάζεται αυτό με την ολοκλήρωση ταυτόχρονα της αγοράς εμπειρογνώμονες για τα κοινωνικά ζητήματα γνωρίζουν καλύτερα από μένα ότι έχουμε ένα περίεργο πλέγμα στην Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι υπεύθυνο και έχει αρμοδιότητες για να χειριστεί το θέμα της ολοκλήρωσης αγοράς, ενώ οι κοινωνικές πολιτικές επαφίονται σε μεγάλο βαθμό στα κράτη-μέλη. Πώς λοιπόν θα φροντίσουμε η διαδικασία της ε, ολοκλήρωσης, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να προχωρήσει και να βαθυθεί, ότι αυτή είναι συμβατή με μια κοινωνική Ευρώπη και μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Δεν πιστεύω ότι τις κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να τις ε, ε, μεταφέρουμε ή να τι εκχωρήσουμε από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό, γιατί έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες και εθνικές παραδόσεις. Οπότε πιστεύω ότι οι περισσότερες ε, κοινωνικές αποφάσεις, ε, οι ανακατανεμητικές, θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό επίπεδο. Δεν θα πρέπει να αναχθούν στο ευρωπαϊκό. Αυτό όμω που θα μπορούσαμε να επανεξετάσουμε είναι η διαδικασία τη ολοκλήρωση τη αγορά. Ώστε όσο προχωρεί να μην έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες, ακούσιες, στις κοινωνικές πτυχές και στις κοινωνικές πολιτικές. Και να σας αναφέρω ένα παράδειγμα που μπορεί να μην είναι το πιο σημαντικό, αλλά σίγουρα είναι από τα πιο επίμαχα. Και κατά τη γνώμη μου, αντί να έχουμε μία εναρμονισμένη ε, επιβεβλημένη άνωθεν κοινωνική πολιτική θα πρέπει να αποφύγουμε η τελειοποίηση της ε, εσωτερικής αγοράς να δημιουργήσει εξαιτία της έλλειψης συντονισμού σε φορολογικά θέματα μία προκατάληψη όλο και μεγαλύτερη κατά του εργατικού δυναμικού και υπέρ του κεφαλαίου και των άλλων παραγωγικών δυνάμεων γιατί οι πιο κινητοί παράγοντες της παραγωγής είναι αυτοί που ε, εποφελούνται περισσότερο από το φορολογικό ανταγωνισμό οπότε, και από την έλλειψη ε, μιας φορολογικής εναρμόνισης, ενός φορολογικού συντονισμού. Πιστεύω ακράδαντα ότι φυσικά εγώ εδώ δέκα χρόνια ασχολήθηκα με το θέμα της εμβάθυνσης, της ολοκλήρωσης της αγοράς και της ε, διασφάλισης της ανταγωνιστικότητάς της. Σε αυτό αφιέρωσα το χρόνο και την ενέργειά μου. Οπότε μην περιμένετε από μένα να πω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ενδοτικοί και να μην είμαστε αρκετά απαιτητικοί σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της αγοράς. Αν όμως αυτή η ολοκλήρωση δεν λάβει υπόψη και τις κοινωνικές συνέπειες, τις κοινωνικές επιπτώσεις, αν οι κοινωνικές επιπτώσεις ε, παραγωνιστούν τελείως ε, από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τότε τα κοινωνικά αιτήματα, οι κοινωνικές αξιώσεις θα μας έρθουν ως μπούμεραγκ. και θα παρεμποδίσουν την απρόσκοπτη ή ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς. Have this as Αυτά είχα υπόψη μου όταν ο πρόεδρος Μπαρόζο, όπως αναφέρατε και εσείς πρόεδρε, ασχολήθηκε με το θέμα της νέας όθησης στην εσωτερική αγορά. Και τους τελευταίους δύο μήνες ε, Είχαμε με πολλές πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαβουλεύσεις και με εταίρους και ειδικέ επιτροπές και έρχομαι σήμερα στη δική σας επιτροπή για να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Έχω τη γνώμη ότι η ενιαία αγορά δεν ε, έτυχε της δέουσας προσοχής ε, υπό το πρίσμα και των ε, παρενεργειών που μπορεί να προκαλέσει σε άλλες πολιτικές. Και μάλιστα ένα απόσπασμα της έκθεσης ΚΟΚ του 2005 που δεν αφορά τη Λισαβόνα αλλά την ενιαία αγορά λέει ότι το πρόγραμμα της ενιαίας αγοράς δεν έλαβε την προτεραιότητα που άξιζε. Αυτό λέει αυτό, λέει ο κύριος Κόκ, είναι ολέθριο ε, πολιτικό σφάλμα, η σφάλμα πολιτικής. Και αυτό το είπε από το 2005, όχι σήμερα, το 2010. Από το 2005 λοιπόν και παρά τις ε, αποφασιστικές ε, και γενικώ επιτυχημένες προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ενιαία αγορά προσέκρουσε σε ενδιασμούς και πριν την κρίση με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Με την κρίση, βλέπε τις α, ε, τάσεις ενός ε, εθνικού προστατευτισμού, αλλά και στη διάρκεια της κρίσης με μία επέλαση της φιλελεύθερης οικονομίας αγοράς. Με αποτέλεσμα η κοινωνική πτυχή να, να, να χάσει την έγκλη αλλά και το φιλελεύθερο μοντέλο το ίδιο. Δεν είναι πολύ ελκυστικό, αλλά θα είναι το μόνο που υπάρχει και θα δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή την οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη. Οπότε θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα αντιμετωπίσουμε το καθένα με τη σειρά του. Γιατί όλες οι χώρες, η μια μετά την άλλη, επιβράδυναν, για να μην πω ότι παρεμπόδισαν τη διαδικασία της ενιαίας αγοράς. Ε, ανακύπτει και το ερώτημα, οι πολίτες απολαμβάνουν τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς. Είναι κοινωνικά φιλική η εσωτερική αγορά. Μήπως ε, θίγει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την απασχόληση. Τι γίνεται με τις εξωτερικές πτυχές της ενιαίας αγοράς. Και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί είναι προβληματισμοί σχετική με την ενιαία αγορά. Πάντως πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μία στρατηγική που απαρτίζεται από δύο τμήματα, άρρηκτα συνδεδεμένα και συμπληρωματικά. Και αυτή θα είναι και η πεμπτουσία των συστάσεων που θα υποβάλω προς τον πρόεδρο Μπαρόζο. Ένα τμήμα της στρατηγικής είναι κάποιες πρωτοβουλίες για την ε, νέα όθηση της ενίας αγοράς, πολλές πρωτοβουλίες και δεύτερη πτυχή εξίσου σημαντική και από άποψη πολιτικού χρονισμού είναι πρωτοβουλίες ώστε αυτή η όθηση της εσωτερικής αγοράς να γίνει κοινωνικώς αποδεκτή, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς που ανέφερα και τις συνησυχίες. Αλλιώς, η αγορά, παρά τους, ε, τις αγαθές προθέσεις και τις βαρύγδουπες διακηρύξεις για την ανάγκη πρόοδου δεν θα σημειώσει ουσιαστική πρόοδο. Πιστεύω ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες, όπως είπε και προηγουμένως, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα πρέπει να αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους αυτή η οδηγία δεν προκάλεσε κεραυνοβόλο έρωτα στην κοινή γνώμη και είδαμε τι διαμαρτυρίες προκάλεσε παντού. Λοιπόν, όλες αυτές τις ανησυχίες θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε, να αφαιρέσουμε τα επίμαχα σημεία και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο δρόμο της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς. Το θέμα της ψηφιακής Ευρώπης επίσης είναι σημαντικό. Πώς μπορεί αυτή η πρόοδο να συντελεστεί, λαμβάνοντα υπόψη όμω και τα συμφέροντα του καταναλωτή και πολλοί άλλοι τομεί. Επειδή όμω εδώ σήμερα επικεντρωνόμαστε στο, στις κοινωνικές πτυχές και με ενδιαφέρουν και οι αντίθετες απόψεις, δεν είμαι πέρα άκρα της εναρμόνισης των κοινωνικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα όμως ένα φορολογικό συντονισμό. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να φοβόμαστε μια συζήτηση για τα θέματα αυτά. Κανένα ζήτημα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν πρέπει να παραμείνει ταμπού. Και με τη συγκρατημένη ισοδοξία κάποιου που το 95-96 ήταν επίτροπος εσωτερικής αγοράς και ανταγωνιστικότητας και έβαλε στο δύο τραπέζι τους 15 τότε υπουργού Εκοφήν και συνεργάστηκε μαζί τους για να καταλήξουμε σε ομόφωνη συμφωνία τον Δεκέμβριο του 1997 για ένα φορολογικό πακέτο που αποτελούσε τη βάση για τη διαδικασία των αποταμιεύσεων, δεδολογικό κώδικα για τη φορολογία των επιχειρήσεων και άλλα. Ήταν μια δέσμη φορολογικών μέτρων. Καμία χώρα δεν ήταν πλήρω ικανοποιημένη με όλα τα στοιχεία του πακέτου του φορολογικού. Αλλά κάθε χώρα βρήκε στο πακέτο αυτό κάτι που την ενδιέφερε, που ήταν ελκυστικό και το εστερνίστηκε. Έτσι μπορούμε με θέματα ενιαίας αγοράς, κοινωνικής πολιτικής, φορολογικής πολιτικής, με όλα αυτά τα στοιχεία μπορούμε να επιχειρήσουμε κάτι παρόμοιο. Ένα θέμα που γνωρίζω καλά και που σας απασχολεί ιδιαίτερα, το αναφέρατε και εσείς κύριε, κύριε Πρόεδρε, και γνωρίζω ότι και η συγγετρία Μπερές ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Τη χρηματοδότηση της κοινωνικής προστασίας του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας μετά την κρίση. Γιατί συνδυάζονται η κοινωνική με τη δημοσιονομική κρίση. Διάβασα ένα άρθρο το περασμένο Ιούνιο στους Financial Times που δεν ήταν και άρθρο κανένα εξωτικού οικονομολόγου, ήταν ενός έγκριτου υπεύθυνου ανθρώπου του Πρωθυπουργού της Φιλανδίας, που έλεγε «Αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ίσω θα πρέπει να αυξήσουμε τη φορολογία τα επόμενα χρόνια, αν δεν θέλουμε απλώ να περικόψουμε δραστικά τις κοινωνικές μας υπηρεσίες προς του συμπολίτες μας. Θέλουμε να αυξήσουμε τη φορολογία με ασυντόνιστο τρόπο και στο βαθμό που χρειάζεται, ώστε να έρθουμε σε αντιπαράθεση, να δημιουργηθεί ένας φορολογικός ανταγωνισμός. Ενώ θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή κατανομή του εισοδήματος και αξιοπρεπή κοινωνική προστασία. Αυτό θα γίνει με ασυντόνιστο τρόπο φίρδιν μίγδιν, οπότε οι κινητοί παράγοντες να υποφεληθούν από αυτό το φορολογικό ανταγωνισμό και να πληγεί το εργατικό δυναμικό. Ή μήπω θα πρέπει να προβούμε σε ένα φορολογικό συντονισμό και σε ένα συντονισμό των πρωτοβουλειών μας. Η έξοδος από την κρίση, το θέμα της, ε, των δημόσιων οικονομικών, ίσως ε, χρήζει ένα νέο βλέμμα για τα θέματα τα φορολογικά. Υπάρχουν κάποια θέματα φορολογικού ανταγωνισμού πραγματικά είναι προβληματικά. Δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο. Αν μπορούσαμε να έχουμε συμμετρικό τρόπο το φορολογικό ανταγωνισμό για τους διάφορες παράγοντες της παραγωγής, εντάξει, μακάρι. Αλλά δυστυχώς ο φορολογικός ανταγωνισμός που ξέρω εγώ είναι σύμμετρος. Και μάλιστα πλήττει αυτούς που θέλουμε να προστατεύσουμε, τους εργαζόμενους. Τι κοινωνική Ευρώπη είναι αυτή που θέλω τυφλή, που γυρίζει την πλάτη στο φαινόμενο αυτό. Πώς μπορούμε μετά να απορούμε και να εξτάμεθα που υπάρχει αντίδραση του κοινού σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση αγοράς, αν το παραμελούμε. Τέλος, δεν μίλησα για την πολιτική ανταγωνισμού. Παρόλο που είναι ακόμη με στην καρδιά μου. Αυτό δεν είναι άμεσα κοινωνικό, αλλά σχετίζεται με την κρίση. Δεν ξέρω αν στα πλαίσια της εντολής σας καλύπτεται και την πολιτική ανταγωνισμού, αλλά προσοχή. Εξετάστε την αμερικανική εμπειρία της δεκαετίας του 30, του πρώτου τμήματος της δεκαετίας του 30, όταν η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει σε παρένθεση τα τους αντιμονοπολιακούς νόμους και να δημιουργήσει καρτέλ όμιλους που ε, από την κυβέρνηση και έκανε επενδύσεις. Αυτό, κατά τη γνώμη των ιστορικών, επιδίνωσε και παρέτεινε την κρίση. Οπότε, μία κρίση δεν σημαίνει θα πρέπει ε, να οδηγήσει σε εγκατάλειψη των αρχών του ανταγωνισμού σε κατάρρευση του ανταγωνισμού. Όταν όμως εξετάζουμε το θέμα του χρονοδιαγράμματος εξόδου από την κρίση, θα πρέπει να κάνουμε μια σημαντική διάκριση. Μπορεί η μακροοικονομική υποστήριξη ε, σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ζήτηση θα μπορούσε να παραμείνει λίγο παραπάνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι και οι μικροοικονομικές ε, ενισχύσεις προς τις βιομηχανίες θα πρέπει και αυτές να διονυστούν. Θέλουμε να συμπαρασταθούμε και ε, να ακούσουμε τον Gains στην κατάσταση αυτή, αλλά να μην ε, κλείσουμε το δρόμο και προχωρήσουμε σε μια δημιουργική καταστροφή. Ευχαριστώ. Θα σας ζητήσω να είσαστε σύντομοι συνάδελφοι, να μην ε, μακρηγορήσετε. Ένα λεπτό. Έχουν ζητήσει ήδη κάποιοι το λόγο. Καταρχάς ο κύριος Τόμας Μαν. Κύριε Μόντι, σας έχουμε ε, ζήσει σαν πολύ επιτυχημένο επίτροπο. Είσαστε κατά της εναρμόνισης ε, και εμείς επίσης η κοινωνική πολιτική είναι θέμα των εθνικών κρατών μελών. Χρειαζόμαστε όμως συντονισμό και νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι γνωστό αυτό που, το τι έχουμε πετύχει. Έχουμε το κοινωνικό ταμείο που είναι το πιο μεγάλο ταμείο. Έχουμε τις μικροπιστώσεις για τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να λάβουν υπό κανονικούς όρους συνθήκες. Έχουμε ε, διοχετεύσει το ευρωπαϊκό Ταμείο παγκοσμιοποίηση προ τι σωστέ ε, κατευθύνσει. Όλα αυτά είναι γνωστά. Ή μήπω ε, θεωρεί ο κόσμος ότι όλα αυτά παραμένουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του, των εθνικών κρατών μελών και δεν είναι γνωστή η ευρωπαϊκή διάσταση. Και γιατί κάνουν τα πανεπιστήμια προ αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πλατφόρμα για την ενημέρωση του κόσμου. Σύμφωνα απόλυτα με την ε, αντίληψη αυτή. Ότι δηλαδή θα πρέπει να αφήσουμε πολλές ε, διοικητικές και κοινωνικές αρμοδιότητες στα εθνικά κρατημέλη. Δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία. Όχι, χρειάζεται πιο πολύ ε, συντονισμός και συγκεκριμένα μέσα κοινοτικά, όπως αναφέρατε το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης και νομίζω ότι έχετε δίκιο. Οι πολίτες δεν ε, γνωρίζουν απαραίτητα τα μέσα αυτά και νομίζω ότι όντως χρειαζόμαστε δράσεις για να κάνουμε πιο ευδιάκριτες ε, τις ε, ενέργειες αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης να σας πω ότι χρειαζόμαστε πέρα από τις θετικές δράσεις και αρνητικές δράσεις, δηλαδή να πούμε σε πολιτικούς, σε εθνικό επίπεδο να σιωπήσουν πια και να δείξουν πιο πολύ προσοχή όταν περιγράφουν τα ευρωπαϊκά μέσα. γιατί όλοι είμαστε εδώ για την πρόοδο των ευρωπαϊκών και εθνικών συστημάτων. Αλλά η αντιμετώπιση των πολιτικών σε εθνικό επίπεδο νομίζω ότι αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Από συντηρητικούς και πάλι η κυρία Χολουμαϊρ. Ähm, Κύριε Μόντι, συμφωνώ με την ε, εκτίμησή σας για την ε, οικονομία της αγοράς, η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη και κοινωνικούς παράγοντες. Και θα ήθελα να σας θέσω την εξή ερώτηση. Μιλήσατε για τον φορολογικό ανταγωνισμό και για την ανάγκη να αυξηθούν οι φόροι επειδή είναι πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις και οι σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών σε ό,τι αφορά τις εισφορές και τις φορολογίας. Θεωρώ, και γι' αυτό σας θέτω και το ερώτημα αυτό, ότι πρόκειται ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να δοθεί σε τα, στα άτομα αυτά που φορολογούνται πολύ χαμηλά, που έχουν πολύ χαμηλές εισφορές. γιατί οι υψηλόμιστοι αυτοί που ε, καταβάλουν υψηλούς ε, φόρους πλήττονται από, τους, ε, από την κατάσταση αυτή και βλέπουμε ότι υπάρχουν μετακαταστάσεις επιχειρήσεων για λόγους φορολογικούς. Κατά δεύτερον, στο πλαίσιο αυτό δεν θεωρείται ότι υπάρχει περιθώριο και δεν θα έπρεπε να συζητήσουμε το φορολογικό dumping όχι μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά και στο εξωτερικό της. Και διαπιστώνω ότι σε πολλές περιπτώσεις λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν ιδιαίτερα α, την μέση τάξη, τις ε, μεσές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ε, κοινωνίας και αυτό ακριβώς στο αυτή ακριβώς το επίπεδο ε, επηρεάζουν αυτές οι αποφάσεις. Λοιπόν, μήπως θα έπρεπε οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνουν υπόψη πιο πολύ αυτή τη μεσαία τάξη. Απάντηση. Θα προσπαθήσω και εγώ, Πρόεδρε, να είμαι πιο σύντομος για τα θέματα φορολογίας. Στα θέματα φορολογίας θεωρούμε ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά τον φορολογικό ανταγωνισμό, γιατί αυτό, ε, αν θέλετε, περιορίζει κάπως τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό που είπατε για το φορολογικό dumping είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και να σας πω ότι υπάρχουν χώρες μεταξύ των νέων κρατών μελών που έχουν παίξει το χαρτί του πολύ χαμηλού ή του μηδενικού φορολογικού συντελεστή για τις εταιρείε. Αλλά και πάλι η κρίση αλλάζει κάπως τις νοοτροπίες. Αναρωτιούνται οι χώρες αυτές μήπως αυτή η τακτική οδήγησε εν μέρη στην κρίση. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ίσως χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη να είναι έτοιμες και πρόθυμες πλέον να εξετάσουν μια λιγότερο επιθετική φορολογική πολιτική, αν παράλληλα θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα για τις ε, εργασίες και καλύτερη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προς τα παλαιά κράτη-μέλη. Αυτό αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα, μία σκέψη, αν θέλετε, για την μεσαία τάξη τώρα, για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά φυσικά συμφωνώ ότι αποτελούν το σκελετό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε απλοποίηση, ναι, αλλά και πολιτική ανταγωνισμού, γιατί πιο πολλές δράσεις του πολιτικής, ανταγωνισμού, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ε, αποτελούν ε, δράσεις χωρίς ε, τακτική, χωρίς πολιτική. Αποτελούν συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες είναι και σκόπιμες. Και να περνάσουμε τώρα στους σοσιαλιστές, να ακούσουμε και τις δύο ερωτήσεις πρώτα. Η κυρία Φερέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η παρουσίαση που ακούσαμε αποδεικνύει ότι καμιά φορά οι κρίσεις δημιουργούν ευκαιρίες. Η Ευρώπη χρειαζόταν να αναζωογονήσει και να αναθεωρήσει το σκεπτικό της, τη φιλοσοφία της. Το γεγονός λοιπόν ότι τώρα αναζητούμε τρόπους για να κάνουμε πιο λειτουργική την εσωτερική αγορά μου φαίνεται μια καλή μεθόδος προσαρμογής. Είχα ερώτηση τώρα για την εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία θα πρέπει να αναθεωρήσουμε, την εξωτερική της δηλαδή πολιτική και έπειτα για τους φόρους. Αναπτύξατε κάποιες ε, παρατηρήσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε και επίσης για τις οριζόντιες πολιτικές δεν θα πρέπει να τις αναπτύξουμε περαιτέρω και σε αυτή την προοπτική και με τι προπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό ως μια πνευματική άσκηση, να ξανασκεφτούμε κάποια στοιχεία της Ευρώπης με την ευκαιρία της κρίσης αυτής, την οποία ακριβώς ως τέτοια θα πρέπει να τη δούμε. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να σταθώ στο θέμα της θενατικής πρόκλησης, την οποία και εσείς αναφέρατε για να ακούσουμε την συμβολή σας. Όπως θα θυμάστε στην οξύτερη περίοδο της κρίσης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικές μορφές ακούστηκαν σενάρια προστατευτισμού με διάφορες εικόνες και σκηνικά να περιγράφονται και να γίνονται και να προτείνονται αλλά αυτά ήταν καρποί φόβων και ανασφάλειας και συνέπεια μια αδύναμη ακόμη νοοτροπία για την εσωτερική αγορά που είναι ρυθμισμένη τώρα. Η απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο και η Επιτροπή να αφήσουν τα κράτη-μέλη επί τη ουσία να διαχειρίζονται από μόνα του την κρίση, όλα αυτά συνέβαλαν στην νέα ανάδυση των αρνητικών αυτών τάσεων. Φαίνεται όμως ότι δεν υπήρχαν μόνο τάσει προστατευτισμού. ως αντίδραση ή ως ενέργεια στα πλαίσια της ε, αγοράς αυτής, της εσωτερικής αγοράς. Υπήρχαν και άλλα προβλήματα που προέρχονταν από τις ε, δυσκολίες της προστασίας αγοράς εργασίας και της αγοράς των επιχειρήσεων. Και εκεί ακούστηκαν ιδέες για φορολογικές πολιτικές οι οποίες και αυτές αντί να συντονίζονται τελικά, περισσότερο ασχολούνται με τα τοπικά συμφέροντα και προτεραιότητες. Αυτό όμω δεν είναι αποτελεσματικό, για να μην πω αντιπαραγωγικό για μια ευρωπαϊκή πολιτική. Το θέμα είναι λοιπόν τι θα γίνει με την προσαρμογή και τη πολιτική ανταγωνισμού. Συνάδελφε, την ερώτησή σας να ακούσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Θέλαμε, κύριε Μόντι, να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτήν την ιδέα τα όσα σχεδίασε το Συμβούλιο ε, και κατά πόσον οι νέες προτάσεις της Επιτροπής δεν ε, εμποδίζουν την αναζωγόνηση της πολιτικής ανταγωνισμού. Ε, του, του Mrs. Στην κυρία Φερέιρα να πω ότι πράγματι πρέπει να αναζωογονήσουμε τη φιλοσοφία μας. Αναφέρατε πρώτη την εξωτερική διάσταση. Στις διαβουλεύσεις μου με τις κυβερνήσεις των κρατών φαίνεται ότι το θέμα αυτό λαμβάνει ένα και περισσότερη σημασία. Ιδίω σε μια περίοδο όπου στην παγκόσμια αγορά βλέπουμε οι Ηνωμένε Πολιτείες να έχουν θετήσει πρόσφατα μέτρα που φαίνονται να είναι χαοτικού σοσιαλισμού βέβαια στην τάση τους, αλλά παραμένουν πιστοί και, και ε, άλλοι παραμένουν πιστοί στις ορθόδοξες αρχές της αγοράς. Εμάς η ολοκλήρωση της αγοράς μας βασίζεται στις αρχές της αγοράς. Θα ήταν καταστροφικό να εγκαταλείψουμε τον έλεγχο των κρατικών βοηθειών ε, ολοσχερός λόγου Αλλά θα πρέπει και όλας να προβάλλουμε την ανάπτυξή μας και τις εξωτερικές μας επιρροές λίγο πιο αποτελεσματικά, ώστε να προβλέψουμε παρόμοιες αρχές, ισοδύναμες αρχές, στο κατάλογο με τους κανόνες μας και σε ένα διεθνές πλαίσιο. Επίσης ζητήσατε περισσότερα σχόλια για τη φορολογική πολιτική. Βλέπω σε πρώτη φάση να υπάρχουν πολλές πτυχές της φορολογικής πολιτικής οι οποίε ζητώνται από τις ίδιε τις επιχειρήσεις... τον επιχειρηματικό κόσμο, για πιο αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της αγοράς. Και από την άποψη των πολιτών όμως. Υπάρχουν πολλοί φορολογικοί φραγμοί για να υπάρχει μια ανετότερη κινητικότητα των πολιτών και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να μην είναι αντιφατικά μεταξύ τους εφόσον δεν προκαλούν και διαφωνίες. Και μετά υπάρχει και η διάκριση μεταξύ κεφαλαίου και αγορά εργασία, όπω είπα προηγουμένω. Λοιπόν, αν τα θέματα όλα αυτά συνεξεταστούν, μπορεί να επιτελεστεί πρόοδο και με μεγάλη χαρά διαπίστωσα ότι στι συμπληρωματικέ του απαντήσει, γραπτέ απαντήσει μετά την ακρόαση, ο υποψήφιο επίτροπο ΕΜΕΤΑ αναφέρει την ιδέα που ήταν ε, κίνητρο για το φορολογικό πακέτο του 1997 να έχουμε ένα φορολογικό φόρουμ με προσώπους από την Υπουργεία Οικονομικών, ώστε να δώσουμε νέα όθηση για να δουλέψουμε πάλι για τη φορολογική πολιτική της Ευρώπης από κοινού. Η πρόταση αυτή είναι πολύ εύστοχη. Η ομάδα αυτή όμως θα πρέπει να προεδρεύεται από την Επιτροπή και όχι νομίζω από κάποια εναλλασσόμενη προεδρία ή από ένα σύστημα κυλιόμενο των κρατών μελών. Πάντως, ε, νομίζω η κρίση θα πρέπει να μας οθήσει να αναθεωρήσουμε και την διάκριση των αρμοδιοτήτων. Εξ όσων εγώ καταλαβαίνω, η, κράτης, η κρίση ε, μας υποδεικνύει μια, έναν υψηλότερο βαθμό κεντρικής αντιμετώπισης κάποιων λειτουργιών όπως των ελέγχων της επίβλεψης, αλλά θα πρέπει να μας ενθαρρύνει και όλα η κρίση να φροντίσουμε να κάνουμε κατανομή των αρμοδιοτήτων βάσει μιας ε, βασικής διαδικτύωσης. Στα πλαίσια της πολιτικής ανταγωνισμού, η μεταρρύθμιση που προτείναμε με, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού βλέπουμε να λειτουργεί καλά. Όμως οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν ενισχυθεί σε σχέση με την κεντρική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Και αυτό είναι θετικό. Μπορούμε λοιπόν στην κοινή γνώμη να προβάλλουμε κάποια έμφαση που δίνουμε σε κεντρικές λειτουργίες για να φανεί ότι δεν αναζητούμε κάποιο μονοπόλιο. Κύριε Κομφεράτη, θα περάσω στα Ιταλικά για λίγο να επιτρέπετε. Εάν θυμάμαι ακόμα την ωραία μου γλώσσα καλά, Συμμερίζομαι απολύτως την άποψή σας για τους προστατευτισμούς και τις βαθύτερες αιτίε τους. Αλλά είμαι λιγότερο επικριτικός από εσάς όταν λέγατε ότι η θέση του Συμβουλίου άφησε τα κράτη-μέλη ελεύθερα να διαχειριστούν όπως νομίζουν την κρίση. Δεν πιστεύω ότι έτσι ακριβώς έγινε. Με όθηση της Γαλλικής Προεδρίας, με το έργο της Επιτροπής, οι ε, πιο ανησυχητικές ε, καταστρεπτικές συνέπειες των κρίσεων στα εθνικά συστήματα και τα γειτονικά τους ε, αναχαιτίστηκαν. Πολλά κρατικά συστήματα διορθώθηκαν χάρη στην παρέμβαση της Επιτροπής. Βεβαίως, ένα από τα διδάγματα της κρίσης και για σας και για μας είναι ότι τίθενται προβλήματα όπως ότι δεν γίνεται να έχουμε μια πολιτική συγκυριακή στην Ευρώπη αποτελεσματική με έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό που είναι τόσο χαμηλό ως, με, χαμηλός ως προς το ΑΕΠ εσωτερικά και σε σύγκριση πάντοτε με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Κύριε Κομφεράτη, με τη δική σας την πολιτική γνώση και τις θεωρητικές σας γνώσεις επίσης, μιλήσατε κατά τη, των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και απευθύνατε μια έκκληση γι' αυτό. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα πολιτικού χαρακτήρα. Στο έργο που κάνουμε με, σε συνεργασία με τον πρόεδρο Μπαρόζο είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε νέες και σταθερές ε, θεωρητικές βάσεις ε, στις αρχές της αγοράς για όλη την Ευρώπη φροντίζοντας οι γενικές παράπλευρες συνέπειες της κρίσης να αντιμετωπίζονται από κοινού. Κάποια στοιχεία που ενίοτε τα αφήνουμε στα χέρια των κρατών μελών να τα επιλύσουν. Έχουμε ακόμα 6-7 ομιλητές, αλλά θα κλείσω τον κατάλογο των ε, ομιλητών και παρακαλώ τους συναδέλφους να τηρήσουν το χρονικό όριο του ενός λεπτού, γιατί δεν θα προλάβουμε. Να κάνω μια ερώτηση εξ ονόματος της Άλντε. Σύμφωνο ότι η ενσωμάτωση κοινοποίηση της αγοράς αποτελεί ένα θέμα ευρωπαϊκό, αλλά ότι τα θέματα αυτά παραμένουν εθνική αρμοδιότητα. Χρειαζόμαστε όμως πιο ευέλικτες αγορές. Με τέτοια τα νέα μέσα όπως το Flex Security, η ευέλικτη ασφάλεια, θα πρέπει να πετύχουμε την προώθηση της αγοράς και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν οι πολίτες συνειδητοποιήσουν ότι συμπεριλαμβάνονται και τα κοινωνικά τους δικαιώματα, δηλαδή ότι όταν μεταφέρονται και μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη δεν θα υπόκειται σημαντικά κοινωνικά μειονεκτήματα. Ρωτώ λοιπόν, αυτή την επιταγή των κοινωνικών ε, αρμοδιοτήτων ε, σε εθνικό επίπεδο, μήπως θα έπρεπε να την αναλάβουμε εν μέρη και σε κοινωτικό επίπεδο. Uh, I, really agree with you. Συμφωνώ, Πρόεδρε, ότι η ενοποίηση προαπαιτεί και προϋποθέτει ευέλικτες αγορές, ευέλικτες αγορές εργασίας ιδιαίτερως. Δεν είπατε κάτι τέτοιο, αλλά θεωρώ ότι και οι δύο είμαστε πεπισμένη ότι αυτό αληθεύει ιδιαίτερα και είναι ακόμα πιο έντονο στην ε, ζώνη ενιαίου νομίσματος, γιατί προκειμένου να λειτουργήσει ε, αυτή η ζώνη με άριστο τρόπο, μια προϋπόθεση λοιπόν είναι να υπάρχουν εύρυθμα λειτουργούσες αγορές, το οποίο προϋποθέτει και την κινητικότητα. Και έχετε δίκιο νομίζω πρόκειται για έναν τομέα, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη μεταφορά δικαιωμάτων, όπου εξ ορισμού τα κράτη-μέλη δεν μπορούν μόνο τους να προχωρήσουν. Χρειάζεται συντονισμός. Πιστεύω ότι αν προχωρήσουμε με τις ιδέες που προσπάθησα να σας παρουσιάσω σε ό,τι αφορά την ενίσχυση το, του κλάδου της ε, ενοποίησης της αγοράς, ενώ παράλληλα θα λάβουμε υπόψη και τα κοινωνικά και τις κοινωνικές διαστάσεις ε, της Ευρώπης, χωρίς... Ε, μάλλον θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση του επωνομαζόμενου σκανδιναβικού μοντέλου, γιατί αυτά τα μοντέλα τι κάνουν, τηρούν α, ε, τις αρχές της αγοράς, αλλά δεν παραμελούν και τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τυποποιημένο μοντέλο οικονομικό και κοινωνικό για την Ευρώπη, αλλά βλέπουμε ότι αν θέλουμε η ενοποίηση της αγοράς να λάβει υπόψη και τις κοινωνικές διαστάσεις, αναπόφευκτα ε, θα καταλήξουμε πιο βόρεια παρά ε, προς ε, τον σημερινό. Μάλιστα, έχουμε ακόμα έξι ομιλητές. Ο κύριος Γκίγκολτ, και ähm, κυρία Μόντι, χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Χαιρόμαστε λοιπόν που βρίσκεστε εδώ μαζί σας. Ήταν ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός μεταξύ του έντονου ανταγωνισμού αφενός και αφετέρου ενός κράτους το οποίο ρυθμίζει και νομοθετεί με ενιαίο τρόπο και με την ε, ρύθμιση αυτή αποτρέπει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι λογικά δεν υπάρχει περιθώριο για φορολογικό ανταγωνισμό στο μοντέλο αυτό, όπως δεν υπάρχει περιθώριο και για άνεσα κοινωνικά δικαιώματα σε μια ενιαία αγορά. Γι' αυτό λοιπόν και δαπανούμε ένα μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ μας για κοινωνικά θέματα και αντίστοιχα λαμβάνουμε και μεγάλο ε, ποσοστό από τις κοινωνικές εισφορές. Με ποια λοιπόν μέσα, με ποια εργαλεία θα προσπαθήσετε να διασφαλίσετε ότι οι ανισότητες σε κοινωνικές δαπάνες και κοινωνικές παροχές θα μειωθούν. Ο κύριος Τεγιώμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που κάθε φορά που βλέπω τον ε, καθηγητή Ντεμόντι, Χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω τον κύριο Μόντι και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Τρει ερωτήσεις έχω να κάνω, συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μιλώντας για κοινωνικά δικαιώματα, θα ήθελα να μας πει ο καθηγητής Μόντι αν συμφωνεί με το κίνημα που ζητάει ένα δεσμευτικό μέσο το οποίο θα δεσμεύει και το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε ό,τι αφορά την τήρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Κατά δεύτερον, πώς αντιμετωπίζετε τις υπηρεσίες κοινή ωφέλειας γιατί βλέπουμε ότι στην Ολλανδία στην παρούσα φάση υπάρχουν πολλά προβλήματα στον υγειονομικό κλάδο. Και τρίτη ερώτηση σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνώ απόλυτα που με όσους ε, τονίζουν τη σημασία της, ε, του κλάδου αυτού, αλλά κάνετε στην ε, έκθεσή σας διάκριση μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττεται από την κρίση και μεταξύ των επιχειρήσεων που δεν πλήττονται, γιατί θα είναι σημαντικό να γίνει αυτή η διαφορά. Η κυρία Μπάστες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον κύριο Μόντι για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση των απόψεών του σε σχέση με την κρίση στην εσωτερική αγορά και τις συνέπειες σε κοινωνικό επίπεδο. Ήθελα να θέσω τέσσερα ερωτήματα κάπως συνοπτικά. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρώτον. Γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό μέσο αυτό για την οικονομική συνεργασία και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Τι άποψη έχει ο κύριος Μόντι για αυτό το θέμα. Νομίζετε ότι πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω επιχειρήσει αυτέ και για σκοπό ενίσχυση τη εσωτερική αγορά και για την θέση μα στην διεθνή αγορά. Δεύτερη ερώτηση. Μετά την κρίση βλέπουμε να υπάρχουν όλα ένα αυξανόμενε τάσει προστατευτισμού Πώ γίνεται να καταπολεμηθούν αυτέ οι τάσει, γνωρίζοντα ότι είναι ένα σημαντικό αίτιο αυτό και για κοινωνικέ τρευλώσει. Τρίτο ερώτημα. Ο αποκλεισμό από την οικονομία της αγοράς, έναν εναλλασσόμενο και μεταβαλλόμενο κόσμο όπω ο δικό μα είναι κάτι που δημιουργεί συνθήκες απαράδεκτης φτώχεια. Είμαστε στο έτος καταπολέμησης τη ένδυα και βάσει τη ανάλυσή σα πώ σκοπεύετε αυτό το τόσο επίκαιρο θέμα να το λάβετε υπόψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πώ λοιπόν βλέπετε αυτό το θέμα και τι μέτρα θα προτείνατε για τον αποκλεισμό από την αγορά κάποιων ε, πολιτών, κατά πόσον πιστεύετε ότι μπορεί να καταπολεμηθεί άμεσα και κατά πόσον αυτό δεν θα πρέπει να οδηγεί σε περαιτέρω φτώχεια. Τέταρτη ερώτηση, εσωτερική αγορά. Πώς βλέπετε την αποτίμηση της εσωτερικής αγοράς από τους Ευρωπαίους πολίτες. Βλέπετε να υπάρχουν προστατευτισμοί και τάσεις ε, ιδεολογικής προκατάληψης των πολιτών. Ποια είναι η άποψη σχετικά. Ε, Mr. Ευχαριστώ κύριε Γκίγκολτ. Θυμάμαι τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που ήδη έχουμε κάνει και η παρουσία σας και μόνο παρόλο που σιωπήσατε στο σημείο αυτό μου θυμίζει ότι δεν ανέφερα καμιά φορά τη διάσταση των κλιματικών αλλαγών και της ενέργειας ακόμη. Οπότε και σε εσά και στα υπόλοιπους ακροατές ε, να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για αυτή την παράληψη. Όμως εργάζομαι σιωπηρά, μεν, αλλά σταθερά, για μια νέα προσέγγιση ιδίω προς την φορολόγηση αυτής της τόσο σημαντική διάστασης. Τώρα, τι μέσα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες σε ένα πρότυπο κοινωνική πολιτική Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με μεγαλύτερη προσοχή και βεβαίω θα ανοίξουμε κάποια στιγμή μια σχετική συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι ο ρόλος των φορολογικών πολιτικών γενικά, και αναφέρομαι και στα μεμονωμένα κράτη-μέλη, θα πρέπει να αναθεωρηθεί εκ βάθρων τρεχόμενα χρόνια. Εδώ κλείνουμε μια εικοσαετία ε, μια κυρίαρχης ιδεολογίας και έτσι θα την ονόμαζα, θα την αποκαλούσα παρόλο που πάντοτε πίστευα ιδιαίτερα στην φιλοσοφία της αγοράς. Μια ιδεολογία λοιπόν που κυριαρχούσε και όπου οι φόροι είναι κακοί και η προοδευτικότητα των φόρων ήταν ε, κάτι αρνητικό. Και πολλές άλλες ε, παρελκόμενες ιδέες. Θυμάμαι το 2004, όταν ήμουν ακόμη επίτροπος, αλλά επρόκειτο να φύγω από την Επιτροπή, αρνήθηκα πρόταση του Ιταλού Πρωθυπουργού να γίνω υπουργό οικονομικών του. Και αυτό διότι δεν συμφωνούσα με τη δική του με το δικό του πρωταρχικό στόχο. Μείωση των συντελεστών του προσωπικού φόρου. Αυτό έβρισκε ότι δεν είναι συμβατό με τις ανάγκες του προπολογισμού και της κοινωνικής πολιτικής της χώρας εκείνη την περίοδο. Νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε εδώ μια ανανεωμένη θεώρηση του όλου θέματος και ιδίω τις σχέσεις μεταξύ κρατών ε, προσώπων και αγοράς. Εδώ σίγουρα πρέπει να συμπεριληφθεί η διάσταση της φορολογικής πολιτικής. Κύριε Ντεγιούγκ, ακούσαμε προσοχή την παρατήρησή σας για ένα νομικό, δεσμευτικό νομικό μέσο, να δεσμεύει όλους δηλαδή, σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα σε δύο τουλάχιστον επίπεδα. Δεν έχω κάποια έτοιμη απάντηση εδώ, αλλά σίγουρα θα χρειαστούμε κάποιες ε, διασφαλίσεις εδώ αν θέλουμε να επιτελεστεί πρόοδος στην διάσταση της αγοράς για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και μετά την πείρα μου στην υλοποίηση των αρχών αυτών επί πέντε χρόνια ως Επίτροπος πρέπει να πω ότι πρέπει να δούμε πώς θα αποφύγουμε ακραίες καταστάσεις και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή από τη μια η Επιτροπή να θέλει να εξαφανίσει, να εξαλείψει ε, τις υπο... κάποιες βοήθειες για την οικοδόμηση λόγω χάρη μιας πυρήνας σε ένα δημαρχείο, από ένα δημαρχείο που μια δημοτική αρχή και από την άλλη καταπολεμήσουμε και την αιμονή των κρατών μελών με κάποιες επιθετικές τάσεις που διακρίνουν από την πλευρά της ε, Επιτροπής. Θα πρέπει σίγουρα λοιπόν να κάνουμε εδώ ένα καλό ξεσκόνισμα. Ο τομέα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο και θα, όπως θα θυμάστε και μετά την απόφαση Χάλμαρκ μας οδήγησε μαζί με την κυρία Κρούς να δημιουργήσουμε ένα σχετικό πακέτο μέτρων. Σίγουρα εκεί πρέπει να γίνουν ακόμη κάποιες διευκρινήσεις, ιδίως ως προς την αναλογικότητα Έτσι θα απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα της κυρίας Μπάστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς πρέπει να ενισχυθεί αυτή η σημαντική συνιστόσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Νομίζω σημαντικό εδώ είναι να θυμόμαστε ότι η ενιαία αγορά πρέπει να γίνει πιο φιλική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περισσότερο να διευκολύνουμε την υποβολή προσφυγών την ταχεία ε, εξέταση των προσφυγών, την εκδίκαση των προσφυγών από τις μικρομεσαίε επιχειρήσει ή τις ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διότι κάποιες φορές από μεγάλου ομίλου ή κράτη βλέπουν να παραβιάζονται τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά. Ουσιαστικά αναφέρατε ένα θέμα τεράστιο και με ρωτήσατε ποιε είναι οι απόψει μου για την καταπολέμηση τη φτώχεια. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε σαφώ ε, λεπτομερέστερα κάποια στιγμή, αλλά το θέσατε το θέμα με μεγάλη ακρίβεια και ευστοχία. Δηλαδή, πώ να βεβαιωθούμε ότι η διεύρυνση τη ε, οικονομία τη αγορά δεν θα οδηγήσει σε απαράδεκτα επίπεδα φτώχεια κάποιου πολίτε. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Όχι μόνο γιατί μα απασχολεί η ευημερία και η σωστή ε, κατανομή του πλούτου, αλλά και ε, για λόγους ε, φιλικής προσέγγισης της αγοράς δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε τις κοινωνικές πτυχές. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε λοιπόν για την πρόσβαση των πολιτών στην ενιαία αγορά προκειμένου να μην φανεί εχθρική αυτή στους πολίτες. Εδώ να θυμίσω στους πολίτες ότι η έκθεση Λαμασούρ μου φάνηκε ιδιαίτερα εύστοχη εδώ που ζητήθηκε, όπως ζητήθηκε από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, αλλά δυστυχώς υλοποιήθηκε σε μηδενικά ποσοστά. Όμως, δεν ήταν καθόλου κακή ιδέα να σκεφτούμε ως βάση εργασίας μας αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Μόντι. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το κατάλογο ομιλητών. Θα είμαστε αναγενείς προς τους επόμενους ομιλητές. Υπόσχομαι στους τρεις συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο ότι θα πάρουν το λόγο στον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Και οι τρεις είναι από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Αλλά ήδη έχουν εκπροσωπηθεί επαρκώς οι σοσιαλδημοκράτες. Ναι, να σας πω το εξής. Αλλά όταν δεν τηρούν οι συνάδελφοι τις χρονικές ε, προθεσμίες τους, τι να κάνουμε. Δεν ζήτησε το λόγο. Δεν ζήτησε το λόγο. Λυπάμαι, λυπάμαι. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα και έχουμε μετά χρόνο για να κάνουμε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι πραγματικά ε, ε, προβλεπόταν στο πρόγραμμα να τελειώσουμε στις 10, έχει πάει 10 και 4 η ώρα. Περβάντς, θα σου δώσω το λόγο ούτως ή άλλως μετά. Δεν έχουμε ερώτηση, χρόνο για ερώτηση. Μπορείς να κάνεις μια μικρή τοποθέτηση όμως αν θέλεις. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, λυπάμαι που δεν θα προλάβετε να απαντήσετε. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε όλο το κύρο σας και να καταλήξετε σε ισχυρά συμπεράσματα. Γιατί αν ε, περιοριστούμε στη λογική ότι η εσωτερική αγορά θα καταλήξει αυτόματα σε κοινωνική εναρμόνιση, θα τα καταφέρουμε. Θα πρέπει να κρατήσουμε τη λογική της εσωτερικής αγοράς. Συμφωνώ με αυτή την αφετηρία. Και όντως στη δεκαετία του 30 ε, οι Αμερικανοί έλαβαν κακές αποφάσεις, αλλά και ο Ρούσβελ το 35 το ίδιο, γιατί παρά ήταν ε, ταχεία η στρατηγική εξόδου. Αν όμως εφαρμόσουμε την πολιτική ανταγωνισμού αμετάβλητη, ενώ οι συνθήκες ανταγωνισμού έχουν αλλάξει ριζικά από την υποκοσμιοποίηση, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αντιληπτή την εσωτερική αγορά στους πολίτες μας και να την αποδεχθούν. Τώρα για τα κοινωνικά ζητήματα. Όλοι συμφωνούσαμε ανέκαθεν με τον Ζακ Ντελόρ ότι η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει ιδιωτική, ε, εθνική αρμοδιότητα. Αλλά δεν θα πρέπει να εμένουμε σε αυτή τη διάκριση μεταξύ της λογικής της ε, ε, εσωτερικής αγοράς που αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ε, κοινωνική πολιτική που αποτελούν τη βάση για τον ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων. Κύριε Μόντι, θα μπορούσατε να είστε ακόμη πιο τολμηρός και φιλόδοξος στις προτάσεις σας. Αν δεν το πείτε εσείς, ποιος θα το πει. Θα έχετε τις προτάσεις σας όπως είχαμε και τις προτάσεις του Ζακ Ντελαροζιέρ θα είναι το σημείο αφετηρίας, αλλά μετά θα αρχίσουν να, να αμβλύνονται. Αν από την αρχή δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι, δεν θα απομείνει τίποτα στο τέλος. Θα βάζουμε συνέχεια νερό στο κρασί μας. Θα πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπιστεί και το φορολογικό και το κοινωνικό ζήτημα. Βρισκόμαστε σε μια οριακή στιγμή, ιστορική. Όχι μόνο για τα φορολογικά, όπως είπατε, αλλά και για τα κοινωνικά θέματα. Και το να απευθεθούμε στην ευφία των κρατών μελών με πολύ δυσίωνες βραχυπρόθεσμες προοπτικές δεν μας αρκεί. Θα πρέπει να βρούμε κάποια εργαλεία, όχι για πλήρη εναρμόνιση των πάντων, αλλά για τη συμπερίληψη κάποιων κοινωνικών κριτήριων. Έχουμε σύμφωνο σταθερότητα, έχουμε μηχανισμού συντονισμού, αλλά χωρί κοινωνικά στοιχεία. Ο Ζακ Δελόρη θέλει τότε να τα συμπεριλάβει. Σήμερα ήρθε η ιστορική στιγμή να το επιτύχουμε. Ελπίζω στην έκθεσή σας να το τονίσετε, γιατί υπάρχουν τρεις πυλώνες. Συνθήκη της Ρώμης, συνθήκη του Μάστριχτ, συνθήκη της Λισαβόνας. Συμφωνώ απόλυτα. Στη συνθήκη της Ρώμης είχαμε την πολιτική ανταγωνισμού. Στη συνθήκη του Μάστριχτ το σύμφωνο σταθερότητας και όλους τους μηχανισμούς της κεντρικής τράπεζας κτλ. Τι έχουμε όμως με τη συνθήκη της Λισαβόνα. Θα περιμένουμε από το Μόντι την απάντηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μόντι που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και σας αποχαιρετούμε. Oh, Äh, Συνάδελφοι, να προχωρήσουμε τώρα και να περάσουμε στο επόμενο πάνελ της σημερινής μας ακρόασης. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς ε, ομιλητές μαζί μας σήμερα. Την εισαγωγή στο θέμα ανεργία και το κοινωνικό κράτος θα μας την ε, κάνει ο κύριος Σερ Τόνι Άτκινσον, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ε, για τα οικονομικά και ήταν σύμβουλος και σύμβουλος του Γάλλου Πρωθυπουργού. Οι άλλοι δύο ομιλητές είναι η κυρία Άλες Κουεντραούγκο, η οποία έχει εργαστεί για τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας επί πολλά χρόνια στην Αφρική και έχει κάνει πολλές δημοσιεύσεις για θέματα εργασιακά, εργατικής ε, νομοθεσίας και για την ε, εργασία των παιδιών. Και τέλος έχουμε και τον κύριο Τζέρεμι Σμιθ, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών από το 2003. Τρεις εμπειρογνώμονες λοιπόν στον κλάδο τους με πολλές ε, δημοσιεύσεις Έχετε τα βιογραφικά τους, δεν πρόκειται να αναφέρω λεπτομέρειες. Και έχετε και τα άλλα έγγραφα για τις εισηγήσεις τους. Να καλέσω λοιπόν τον κύριο Sir Tony Atkinson να κάνει την εισαγωγή. Έχει 12 λεπτά στη διάθεσή του, επειδή κάνει και την εισαγωγή ακριβώς, και οι υπόλοιποι 8 λεπτά. Thank you very much uh, for inviting me. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια και ο καθηγητής Μόντι μίλησε για τα μονοπόλια, θα σας πω, παρόλο που αναφέρεται με καθηγητής στα πανεπιστήμια του Oxford, του Cambridge και του Harvard, στην πραγματικότητα είμαι καθηγητής μόνο στο Oxford. Αλλιώς ε, θα καταλάβανα πολλές από τις σπάνιες θέσεις εργασίας που ήδη υπάρχουν, αν ήμουν πολυθεσίτης. Η δική μου ομιλία είναι η φυσική συνέχεια της προηγούμενης ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε με τον κύριο Μόντι. Τόνισε την διάκριση μεταξύ της ανάγκης ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ε, αφενός και αφετέρου των κοινωνικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να την συνοδεύουν αφετέρου. Εγώ ακριβώς ε, για το ίδιο χάσμα θα μιλήσω, θα μιλήσω αλλά σε μακροοικονομικό επίπεδο. Φαίνεται ότι υπάρχει μία ρήξη στην συζήτηση που γίνεται μεταξύ της κοινή γνώμης αφενός και των ακαδημαϊκών κύκλων αφετέρου. Οι συζητήσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο για την ε, πτώση του ΑΕΠ, μακροοικονομικές ανισορροπίες, ε, έλλειμμα, χρέος, χρηματοοικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα συζητούνται από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά έχουμε τα προβλήματα στα νοικοκυριά, την πτώση του εισοδήματο, το βιωτικό επίπεδο και τις μελλοντικέ προοπτικές. Την εβδομάδα αυτή συμμετείχα σε δύο συνεδριάσεις, μία από τη Γενική Διεύθυνση έρευνα για τις ε, κοινωνικές ανισότητες στην Ευρώπη και την επόμενη μέρα ήμουν σε μία συνεδρίαση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου για την έξοδο από το υψηλό δημόσιο χρέος. Και αυτό που με άφησε άναυδο είναι ότι οι δύο αυτές συζητήσει γίνονταν τελείω ε, ε, απομονωμένα και ξεκομμένα μεταξύ τους. Υπάρχει μεγάλο ρήγμα, λοιπόν. Επίσης έχουμε όλα αυτά τα μέτρα για τα φορολογικά ζητήματα που όμως έχουν σοβαρές επιπτώσεις ε, στις βιωτικές συνθήκες των ανθρώπων, των οικοκυριών, των οικογενειών. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που έχουμε για αυτή τη συζήτηση και την ακρόαση και σας συγχαίρω που την οργανώσετε. Θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Προσπάθησα να σκεγγραφήσω τα πράγματα με απλό τρόπο. Μερικά από τα στοιχεία ε, της ε, ευρύτερης μακροοικονομίας και πώς επηρεάστηκε από την ύφεση αυτή την ύφεση που αποτέλεσε τη φυσική απόρρεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Είχαμε πολλά διαδοχικά στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν αυτό που λέμε τη, τη μετά το Λέμαν, τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ο κόσμος διαπίστωσε ότι τα χρήματα που είχε ήταν πολύ λιγότερα, το σύστημα κατέρευσε, χρειάστηκε να εισέλθουν οι κυβερνήσεις για υποστήριξη και φτάσαμε στο δεύτερο στάδιο, τη συνέπεια στην πραγματική οικονομία. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ε, αύξηση της ανεργίας. Αλλά δεν είχαμε μόνο ανεργία, είχαμε μειωμένη απασχόληση, μισθολογική πίεση στην αγορά εργασίας και στο, στην κεφαλαία αγορά ε, λιγότερα κέρδη και μείωση των φορολογικών εισοδημάτων σε ε, κρατικό επίπεδο. Και οι αυτόματοι σταθεροποιητές δυστυχώς δεν επιτέλεσαν το ρόλο τους. Αυτό είναι το στάδιο που βρισκόμαστε. Αλλά αυτό που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο είναι τι μέλη γενέστε. Ποιο είναι το τρίτο στάδιο. Το τρίτο στάδιο είναι εκεί που θα βιώσουμε τις συνέπειες που κατά πάσα πιθανότητα δυστυχώς θα ξεπεράσουν τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής αστητείας. Και δεν μιλάω μόνο για το δημόσιο χρέος που θα παραταθεί, αλλά οι άνθρωποι, οι συμπολίτε μας ε, θα εξακολουθούν να νιώθουν στο πετσί τους τα παρατεταμένα αποτελέσματα αυτής της, χρήσης, της κρίσης. Ιδιαίτερα ε, οι νέοι, αυτοί που τώρα μπαίνουν στην αγορά εργασίας ή μόλις μπήκαν, θα νιώσουν αυτές τις συνέπειες και στο μέλλον και στις, ε, στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και στις απολαβές τους. Επίσης και στην κεφαλαία αγορά θα παραμείνουν τα αποτελέσματα. Γιατί όσοι έκαναν αποταμιεύσει και οικονομίες για τα γεράματά τους θα ε, βιώσουν για πολύ καιρό ακόμη αυτή την ανασφάλεια και θα σταθούν ίσως ότι δεν μπορούν να προβλέψουν για το μέλλον όπως θα ήθελαν ούτε οι οικονομίες τους θα έχουν το αναμενόμενο στήριγμα. Το πρώτο προφανές σημείο που δεν περιλαμβάνεται καν στις διαφάνειες, αλλά είναι αυτονόητο, είναι ότι θα περάσει αρκετός καιρός για να συνειδητοποιήσουμε το εύρος. Πρόσφατα είχαμε τις, τα τελευταία στοιχεία για το Βρετανικό ΑΕΠ για, πέρυσι, το, για το τελευταίο περσινό τρίμηνο Έχουμε για αυτά πληροφορίες, αλλά ελάχιστα γνωρίζουμε για το τι γίνεται σε επίπεδο νοικοκυριών. Για παράδειγμα, το επίπεδο φτώχειας που μας έδωσε η Eurostat για το 2008 αφορά το οικογενειακό εισόδημα για το 2007. Δηλαδή, έχουμε δύο-τρία χρόνια απόσταση. Γιατί το 2010 που υποτίθεται είναι Ευρωπαϊκό Έτο Καταπολέμηση Φτώχεια και Κοινωνικού Αποκλεισμού, στηρίζεται ουσιαστικά σε στοιχεία εισοδήματο του 2007. Θέλουμε μια επικαιροποίηση των στατιστικών μα στοιχείων για να έχουμε παρακολούθηση τη πορεία του βιωτικού επίπεδου ε, πρόσφατη και όχι του παρελθόντος. Επίσης, θα πρέπει από την αρχή, εξάντεκ των προτέρων, να διαρωτηθούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, η επιπτώσεις αυτής της κρίσης στα άτομα, στις οικογένειες και να δούμε αν μπορούμε να διδαχθούμε και από το παρελθόν. Αυτά τα σημεία θα με απασχολήσουν στον υπόλοιπο μου χρόνο. Ποιες εξελίξεις αναμένουμε. Πριν από ένα χρόνο είχα προτείνει και βλέπω ότι μ' άκουσαν η Επιτροπή, όσα και άλλες οργανώσεις, ότι αυτό που έγινε στη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να γίνει και στα κοινωνικά ιδρύματα. Δηλαδή, να διαρωτηθούμε πώς και τα κοινωνικά ιδρύματα θα επιβιώσουν από την κρίση. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και εξάντε. Γιατί έχουμε πολλές διατάξεις και πρόνοια για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την ύφεση. Έχουμε για παράδειγμα επιδόματα ανεργίας, ε, ασθένειας, αναπηρικές άδειες. Έχουμε προστασία εισοδήματος για όσους έχουν χάσει τις οικονομίες τους. Υπάρχει δυνατότητα στήριξης αυτών. Επίσης, όλο και περισσότεροι έχουν κάποια ωφέλη που συνδέονται με το εισόδημά του στην εργασία. Βέβαια, όταν το εισόδημα μειώνεται, μειώνονται και τα συναφή αυτά επιδόματα. Μπορούν όμως μέσα από τον in-work benefits, των επιδομάτων που σχετίζονται των δευτερευόντων ωφελών από το εισόδημα, να μπορούν να υποστηριχθούν. Σήμερα η κατάσταση δεν είναι παρόμοια με αυτή του 1929. Έχουμε κράτος πρόνοιας με τα πολεμικά, που αυτόματα παρέχει ε, ε, βοήθεια, αρρωγή στους ε, πολίτες που βιώνουν μια μείωση του εισοδήματός τους. Επίσης ε, υπάρχουν πολύ σημαντικές δυστυχώς τρύπες, πολύ σημαντικά κενά σε αυτό το δίκτυο ασφαλείας που υπάρχει καταρχήν αλλά στην πράξη μερικές φορές δεν είναι τόσο ορατό. Καταρχήν ποια είναι η κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε από τα στοιχεία ότι οι άνεργοι το 2005 αν τους ρωτούσαμε παίρνετε τα επιδόματα ανεργίας ρώτησε ανθρώπου που ήταν άνεργοι για 4 με 6 μήνε, δηλαδή αρκετό καιρό, όχι μόλι είχα χάσει την απασχόλησή του. Και βλέπουμε ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τρίτο των ανέργων δεν λάμβανε αυτό το επίδομα ανεργία που δικαιούνται. Ήταν χαμηλό σε Αυστρία-Γερμανία, υψηλό στι βαλτικέ χώρε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τι Μεσογειακέ χώρε. το ποσοστό. Δεν ξέρω, ίσως αυτό σχετίζεται επειδή είναι κανείς κοντά στη θάλασσα, σε παραθαλάσσιες περιοχές. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν φτάνει το σύστημα αρρωγής των ανέργων στους δικαιούχους πάντα. Και την περασμένη εβδομάδα η Λεμόντ είχε πηχαίο τίτλο «Ένα εκατομμύριο άνεργοι χάνουν τα δικαιώματά τους από το 2010 και μετά». Δηλαδή το, το ζήτημα επιδεινώνεται. Οπότε θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα δούμε εκ των προτέρων και να δούμε πώς θα λειτουργήσουν αργότερα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, ε, πολλοί δεν λαμβάνουν τα επιδόματα που δικαιούνται. Οπότε δεν είναι βέβαιο ότι το σύστημα κοινωνικής προστασίας μας είναι πραγματικά αποτελεσματικό. Και περνάμε στο, από το εξάντε, από την, εκ των προτέρων πρόβλεψη, στην πραγματική κατάσταση. Και εξετάζουμε κυρίως τους χαμηλούς εισοδηματίες και μετά ε, τα υψηλότερα εισοδήματα. Βέβαια, η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε περίπου στα υψηλά εισοδήματα περισσότερο. Βέβαια, ο κόσμος σήμερα δεν είναι όπως το 1929. Το 1929 και τα υψηλά εισοδήματα επλήγησαν πολύ σοβαρά από την οικονομική κατάρρευση, από το κράχ. Αν δούμε τις ε, πρόσφατες ε, υφέσεις εξαιτίας τραπεζικών κρίσεων, σε όλες και αυτές τις κρίσεις ε, που εντόπισε ο ΣΑ, σε μια πρόσφατη μελέτη, λέει ότι η περίοδος ύφεση είχαμε τα εισοδήματα του, των υψηλότερων εισοδημάτων αυξήθηκαν κατά 1% όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οπότε αυτό που οι πλούσιοι αυτό που οι πλούσιοι αποκαλούν πρόβλημα της φτώχειας, οι φτωχοί αποκαλούν πρόβλημα των πλουσίων. Θα πρέπει να δούμε και τις δύο πτυχές. Να πούμε και δύο λόγια πριν ολοκληρώσω για το πακέτο, το ογκοδέστατο πακέτο που πρότεινε πέρσι ο πρόεδρος Ομπάμα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όχι μόνο θέτησαν ένα τεράστιο πακέτο εναυσμάτων, Και το πρόβλημα της φτώχειας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης σημαντικό. Το πακέτο αυτό θεωρήθηκε ως το κοδέστερο πακέτο υποστήριξης φτώχειας με τα πολεμικά. Και έγινε σχεδόν διακριτικά αυτό το πακέτο. Το παρατάθηκε για παράδειγμα ε, ή επεκτάθηκε το δικαίωμα επιδόματος ενέργειας Και μόνο αυτό το μέτρο είναι πολύ σημαντικό και καλό θα ήταν να το μιμηθούν και πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δίνουν πια επίδομα ανεργία 78 εβδομάδε. Στην ε, Μεγάλη Βρετανία είναι μόνο 26 εβδομάδε η διάρκεια του επιδόματο ανεργία. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα ίσω καλό θα ήταν να το μιμηθούν και πολλέ χώρε μέλη. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω τώρα. Θα πρέπει, αντί να μιλάμε μόνο για πτώση του ΑΕΠ, να εμπλέξουμε και τον κόσμο στην όλη συζήτηση. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης για να γνωρίζουμε τι συνέβη πέρυσι και όχι μόνο πριν από δύο-τρία χρόνια, να δούμε πραγματικά πώς επηρεάστηκε το βιωτικό επίπεδο και αν υπάρχουν εύλογοι λόγοι ανησυχία και βραχυπρόθεσμα σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ανεργίας, αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Πόσες οι επιπτώσεις αυτές για πόσο καιρό θα επηρεάσουν τις βιωτικές συνθήκες του κόσμου. Και το πιο σημαντικό είναι κάτι που επαφίεται στα δικά σας χέρια. Αυτό που θα συμβεί δεν είναι αναπόφευκτο, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις πολιτικές των κρατών μελών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας κάνατε την εισαγωγή στο θέμα αυτό και να δώσω το λόγο πάρα αυτά στην κυρία Κουεντράουγκο. Monsieur le Président de la Commission, euh, euh, Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ήθελα κατά πρώτον να σας ευχαριστήσω που καλέσατε το Περιοδευτήριο Εργασία για να παρακολουθήσει τις συζήτησή σας. Πολύ σύντομα ήθελα να αναπτύξω τρία θέματα. Πρώτα απ' όλα τις συνέπειες της κρίσης στην πραγματική οικονομία. Έπειτα θα σας μιλήσω για τις μεγάλες αδρές γραμμές δράσης που λάβαμε στο ILO, στο Διεθνές Γραφείο για να αντιμετωπίσουμε την κρίση σε συνεργασία με τους εταίρους μας και μετά θέλουμε να δούμε τι θεώρηση έχουμε για το μέλλον στα πλαίσια των εταιρικών σχέσεων που έχουμε διαμορφώσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό και συχνά το αμελούμε όταν μιλάμε για την κρίση στην απασχόληση. Μιλάμε μόνο για ανεργία. Όμως, βάσει του ορισμού της εξωπρεπούς εργασίας, η απασχόληση είναι απλώς μια διάσταση. Υπάρχουν άλλες διαστάσεις που είναι κοινωνική προστασία, τα θεμελιώδη δικαιώματα τη εργασία και όλα αυτά αποτελούν μέρο του κοινωνικού διαλόγου. Όταν ένα από αυτά τα στοιχεία διαταραχθεί, θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση ελλείμματο τη αξιοπρέπους εργασία. Όταν μιλάμε λοιπόν για την κρίση και τι συνέπειε τη κρίση στην απασχόληση, πρέπει να έχουμε σε κάθε περίπτωση κατά νου και αυτές τις άλλες πτυχές, τους άλλους παράγοντες που είναι θεμελιώδεις. Κυρίω γιατί το Διεθνέ θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι αλληλένδετα, δεν μπορούν να διαχωρίζονται ενισχύονται αμοιβαίω και αυτό βάσει μιας δήλωσης που έχουν εγκρίνει όλα τα κάτι μέλη του οργανισμού μας. Μια σταθερή επιβεβαίωση των ε, αξιών που εκφράζουμε ως οργανισμός. Ε, πριν από λίγες μέρες στον Ταβό, ε, ετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε μια σειρά από αριθμούς και στην αίθουσα έχετε και ένα ανακοινωθέν τύπου με τις λεπτομέρειες της έκθεσής μας για τις τάσεις της απασχόλησης παγκοσμίω. Απλώς κάποιους αριθμούς να σας παρουσιάσω για να έχετε μια εικόνα του εύρους του φαινομένου. Ε, ο οργανισμός μας θεωρεί ότι στον κόσμο σήμερα υπάρχουν 212 εκατομμύρια άνεργοι, δηλαδή 34 εκατομμύρια για το έτος 2009. Οι προβλέψεις δεν είναι καθησυχαστικές. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω χάρη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζουμε ότι 3 εκατομμύρια άτομα θα προσθεθούν ε, ποσοστά ενεργείας το 2010 και μόνον. Τι σημαίνουν οι αριθμοί αυτοί. Νομίζω ότι τα αριθμητικά στοιχεία μας θυμίζουν δύο βασικές ιδέες. Πρώτα απ' όλα, πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν πρόσωπα, εκατομμύρια γυναίκες, παιδιά, άντρες, που προοδευτικά ε, φαίνεται σταδιακά περνάνε σε συνθήκες φτώχεια και δεν έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν στην παραγωγή πλούτου. Βρίσκονται λοιπόν στο περιθώριο της κοινωνίας. Η δεύτερη ιδέα είναι ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, να προσέξουμε το στοιχείο αυτό. Επειδή στις εφημερίδες μιλάμε για ανάκαμψη, για έξοδο από την κρίση και την ύφεση. Να μην ξεχνάμε τα διδάγματα του παρελθόντο. Υπάρχει πάντοτε μεγάλη διαφορά μεταξύ τη οικονομική ανάκαμψη και τη ανάκαμψη σε επίπεδο παραγωγή θέσεων εργασία. Μόνο για τι αναπτυσσμένε χώρε οι προβλέψει λένε ότι πριν φτάσουμε σε επίπεδα απασχόληση παρόμοια με αυτά πριν την κρίση, θα πρέπει να περιμένουμε στο 2013. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Επίση, είναι σημαντικό ότι γνωρίζουμε από την πείρα, εκπείρας ότι όταν υπάρχουν ισχυρά συστήματα κοινωνικής προστασίας τα οποία υλοποιούνται αποτελεσματικά, τότε μόνο αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και φτώχεια. Να αναφέρω το πρόγραμμα Welfare Familia στην Βραζιλία, το οποίο κατάφερε να βγάλει από τις συνθήκες φτώχειας 11 εκατομμύρια οικογένειες, δηλαδή 50 εκατομμύρια άτομα, λίγο πολύ. Και οι άλλες παράμετροι της αξιοπρεπούς εργασίας, ο κοινωνικός διάλογος δηλαδή, που επιτρέπει στους εργοδότες και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην διαδικασία λήψη αποφάσεων, να επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό γίνεται μόνο μέσω του κοινωνικού διαλόγου. Το δεύτερο θέμα που ήθελα εδώ να αναπτύξω σύντομα είναι ότι πραγματικά χρειάστηκε να αναπτύξουμε μια νέα φιλοσοφία, ένα νέο σκεπτικό, για να εξετάσουμε τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Πρώτα απ' όλα δώσαμε έμφαση στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους, κάτι που δεν ήταν ε, η πάγια τακτική μας προηγουμένως. Έπειτα, η ανάγκη να ε, μεταρρυθμιστεί το παγκόσμιο οικονομικό αρχιτεκτόνημα είναι πλέον μια επιτακτική ανάγκη και είναι πλέον ε, στον κατάλογο των προτεραιοτήτων μας. Ακόμη είναι σημαντικό ότι διεφάνει αμέσω από την κρίση ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη συνοχή στη δράση μας. Δεν πρέπει ο καθένας να παρεμβαίνει κατά τρόπο άτακτο, αλλά όλοι να ενώσουμε τις προσπάθειε μας και να προσπαθήσουμε να έχουμε κατάλληλες κοινέ αποκρίσεις σε προβλήματα κοινά. Μιλάμε για προβλήματα διεθνών διαστάσεων. Οπότε στην κρίση πρέπει να απαντήσουμε ακριβώς με λύσεις παγκόσμιας διάστασης. Οι εταιρικέ μα σχέσει μα επισημαίνουν και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Η διαδικασία του G20 έδειξε το κύρο τη. Γιατί απάντησε σε προβλήματα τη πραγματική οικονομία και τη απασχόληση ε, προκειμένου να ξεφύγουμε από τι συνθήκε τη παγκόσμια κρίση. Η κρίση έχει πάρα πολλές πτυχέ όμω. Καμία αρχή με τις αρμοδιότητές της μόνη και απομονωμένη δεν μπορεί να την επιλύσει και να την αντιμετωπίσει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας ήταν ο πρώτος οργανισμός που έδωσε μια ξεκάθαρη απόκριση στην κρίση, όσο το δυνατόν συντομότερα. Από τον Νοέμβριο του 2008 δημιουργήθηκε ένα πακέτο μέτρων. Δηλαδή, ένα πάκετ πολιτικών μέτρων που θα επέτρεπε στις χώρες που επιθυμούν να τα υλοποιήσουν για να βγουν από την κρίση μιλάμε για έναν κατάλογο με μέτρα ευέλικτο. Για μέτρα τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους και την αποτελεσματικότητά τους και ήδη εφαρμόζονται από κάποια κράτη. Έχουν δείξει τα μέτρα αυτά τη δυνατότητά, τη δυνατότητά τους να αναχαιτήσουν την κρίση. Έτσι λοιπόν ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας θεωρεί ότι χάρη στο πακέτο κοινωνικών μέτρων που σχεδιάστηκαν ιδίως από τις χώρες του G20 μπορέσαμε να διατηρήσουμε 7-11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον πρέπει να ε, βάλουμε πάλι πρώτη προτεραιότητά μα στην ανάπτυξη. Και εδώ χρειάζεται να ακολουθήσουμε μια διτή προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα, η υλοποίηση του Παγκόσμιου Συμφώνου για την Απασχόληση. Αυτό είναι ένα χάρτη πορεία για τον δικό μα τον οργανισμό. Και επιμένω εδώ στον οργανισμό μα, διότι ο οργανισμό αποτελείται από τα κάτι μελη του, από τι ενώσει εργοδοτών και εργαζομένων. Αυτοί στηρίζουν τον οργανισμό και τον βοηθούν να υλοποιήσει το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Απασχόληση το οποίο σε μεγάλο βαθμό στήριξαν όλα τα θεσμικά όργανα παγκοσμίω συμπεριλαμβανομένου το G20 και το G92. Δηλαδή όλα τα κράτη που συμμετέχουν στον οργανισμό μας και στα ΟΗΕ. Πρόκειται για μια πρόκληση διεθνών διαστάσεων αλλά και μια πρόκληση εθνική. Διότι απευθύνεται στα κράτη, στις κυβερνήσεις το σύμφωνο αυτό αλλά και στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους. Να δώσω εδώ ως παράδειγμα την ανάγκη που έχουν οι επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο τις επιχειρηματικές τους όπως ονομάζονται ευθύνε. Επίσης, ο κοινωνικό διάλογος απέδειξε επανειλημμένος ότι όταν οι εργαζόμενοι και εργοδότε συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τότε υπάρχουν περισσότερε ε, δυνατότητες να απαντήσουν στα πραγματικά προβλήματα γιατί ξέρουν και τι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν στην πράξη. Επίσης, υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση που είναι σημαντική. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το γεγονό ότι τώρα ανακάμπτουμε από την κρίση δεν σημαίνει ότι προοδευτικά μπορούμε να εγκαταλείψουμε όλα αυτά τα εξαιρετικά κοινωνικά μέτρα που αναλάβαμε για να στηρίξουμε του ε, φτωχότερου. Διότι τότε μπορεί να ξαναβρεθούμε σε κατάσταση ακόμη δυσχερέστερη. Υπάρχει προφανώ η ανάγκη να βοηθήσουμε όλε τι χώρε που δεν έχουν τα περιθώρια στον προπολογισμό του ή στην πολιτική του να αναλάβουν μόνοι του μέτρα για να ξεφύγουν από την κρίση. Πρέπει να του δώσουμε ουσιαστική βοήθεια και να καλύψουμε τι ανάγκε του. Το τελευταίο θέμα που ήθελα να αναπτύξω εδώ είναι η εταιρική μα σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια εταιρική σχέση υποδειγματική. Και αυτό απλώ και μόνο διότι οι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινέ με τι δικέ μα. Δεν θα ήθελα να περάσω τώρα στις λεπτομέρειες της στήριξη που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο του ΟΗΕ, αλλά και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τεχνικής συνεργασίας. Είναι σημαντικό εδώ να πούμε κατά κύριο λόγο ότι περάσαμε πολύ κοντά από μια απόλυτη καταστροφή, αλλά καταφέραμε να την αναχαιτήσουμε. Η κρίση αυτή είναι ανθρωπογενεί. Δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε. Και πλήττει του ανθρώπου πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει λοιπόν απλό τρόπο να την ε, δαμάσουμε. Σα ευχαριστώ κυρία μου. Να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Σμίτ. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου επιτρέπετε να θέσω και τις δικές μας ε, απόψεις εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών που είναι μια οργάνωση ομπρέλα που συνενώνει τις εθνικές σχετικές αρχές να πω ότι οι ευρωπαϊκές αρχές ε, είναι πολύ διαφορετικές σε ό,τι αφορά το μέγεθος, τις αρμοδιότητες και τις χρηματοοικονομικούς πόρους τους. Και νομίζω όμως ότι μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν στο σύνολό τους διατραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τους μειονεκτούντες, τους ανέργους, τους κοινωνικά περιθυροποιημένους Περίπου το 10 έως το 25% δαπανούν στις ευρωπαϊκές χώρες για να καταλάβετε ε, ποια είναι η κλίμακα στην οποία δημιουργούν, ε, εργάζονται. Και επίσης ε, σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιακές επενδύσεις, σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, σε πράσινες επενδύσεις, είναι πάρα πολύ ενεργές, αλλά οι αρχές αυτές, όπως και οι τοπικές αρχές, πλήττονται έντονα από την οικονομική κρίση, που ασκεί τεράστια πίεση σε αυτές και επιτάσσει να αναλάβουν τα καθήκοντά τους σε μια δύσκολη εποχή. Και σε πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο, έχουμε κάποια στοιχεία και φυλάδια εδώ, τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους επιδεινώθηκε η κατάσταση κατά 70% και το 2010 στην Σκανδιναβία θεωρούσε ο κόσμος κατά 10% ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Το 50% θεωρούσε ότι θα μειωθούν οι προϋπολογισμοί για κοινωνικά θέματα και άλλοι οι υπόλοιποι πίστευαν ότι θα πάγωναν οι σχετικές χρηματοδοτήσεις και το 60% ότι οι κυβερνητικές μεταφορές στις ε, δημοτικές αρχές είχαν ε, μειωθεί. Και ξέρουμε ότι είχαν αυξηθεί οι πιέσεις ως προς τις ε, δαπάνες. Ο πρόεδρος ε, της Γερμανικής Ένωσης Δήμων παρουσίασε τα εξή. Ε. Η πρόεδρος είπε τον Νοέμβριο ότι τα έσοδα των εμπορικών εισοδημάτων θα έχουν περιοριστεί κατά 20% και η εκχώρηση κονδυλίων στις τοπικές αρχές θα μειωθεί το επόμενο έτος. Οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση αυτή. Μάλλον η κατάσταση θα επιδεινωθεί από τις φορολογικές περικοπές. Και παράλληλα ανεβαίνει το κόστος των κοινωνικών δαπανών, το οποίο είναι αναπόφευκτο κατά την οικονομική κρίση και ούτω καθεξής. Είναι σαφές λοιπόν και αυτό αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα για όλη την Ευρώπη ουσιαστικά. Επίσης ε, φοβούμαστε ότι ο αντίκτυπος των αυξανόμενων ε, ελλημάτων σε εθνικό επίπεδο και των ε, εθνικών χρεών θα μειώσει περαιτέρω τα εισοδήματα σε μια εποχή που η πίεση για την παροχή βοήθειας προς τους ε, ανέργους και τους υποαπασχολούμενους γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Αυτό που θα θέλαμε η Επιτροπή να σημειώσει είναι το εξής. Καταρχάς ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Ευρώπη χρειάζονται ένα περιθώριο ελιγμού αλλά έχουν πιο περιορισμένο περιθώριο από τις εθνικές αρχές και σε κάποιες ε, περιπτώσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν καν σε δανεισμό για να καλύψουν τα κενά στον προϋπολογισμό. Είναι πιο περιορισμένες δηλαδή από ότι οι εθνικές αρχές σε κάποιες περιπτώσεις. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή αυτή θα τονίσει τον ουσιώδη ρόλο των εθνικών και περιφερειακών, των, συγγνώμη, περιφερειακών και δημοτικών αρχών και θα ενθαρρύνει και από πλευράς πολιτικών και τις ευρωπαϊκές αλλά και τις εθνικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα επηρεαστούν δυσανάλογα οι περιφερειακές και οι δημοτικές αρχές γιατί υπάρχει ο κίνδυνος και ο φόβος ότι οι εθνικές αρχές θα θεωρήσουν ότι οι περικοπές είναι πιο απλές σε χαμηλό επίπεδο, σε δημοτικό επίπεδο. Δεν ενισχύει όμως αυτό. Και φοβούμαστε ιδιαίτερα ότι στην παρούσα φάση που η όλη διαδικασία της αποκέντρωσης ε, των υπηρεσιών κινδυνεύει να σταματήσει και να επανέλθει στα χέρια της εθνικής κυβέρνησης, των εθνικών κυβερνήσεων. Όλος παραδόξης, για πρώτη φορά έχουμε μια συνθήκη, τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τονίζει το ρόλο της ε, των τοπικών αρχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά και, τα, και την επικουρικότητα. Θα θέλαμε λοιπόν να τονίσετε ότι υπάρχει ανάγκη να μην αντιστραφεί αυτή η μακροπρόθεσμη διαδικασία δημοκρατικής αποκέντρωσης σε ό,τι αφορά την οικονομία και τις υπηρεσίες, γιατί οι τοπικές αρχές χρειάζονται τις, ε, την το περιθώριο ελιγμού που ξέρουμε ότι θα τους χρειαστεί για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των επόμενο, στα επόμενα χρόνια. Φυσικά έχουν υποστεί τεράστιες πιέσεις τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να βρούμε καινούργιου τρόπους για να παρέχουμε τις υπηρεσίες και τις, ε, το έργο που χρειάζεται. Και συμφωνώ με τον ε, Κύριε Μάρτιν, σε ό,τι ανέφερε για τις ε, υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένε περιπτώσεις έχουν ε, υιοθετήσει στρεβλές προσεγγίσεις ως προς την σχέση των ε, νομοθέσεων εσωτερικής αγοράς και σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος που παρέχονται σε περιφερειακό επίπεδο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το διακοινωτικό επίπεδο. και θεωρούν ότι αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος για να τεθεί και σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο περί Συμβάσεων. Και θα επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριος Μόντι, ότι σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται ε, απόπειρα να εμπλακεί κανείς και σε πράγματα τόσο απλά όσο η χρηματοδότηση μιας ε, δημοτικής πισίνας, για παράδειγμα. Άρα στρεφόμαστε προς εσάς για να μας βοηθήσετε επ' αυτών των θεμάτων, θεμάτων αυτονομίας και να επιτρέψουμε αυτό που η Επιτροπή των Περιφερειών ε, πρόσφατα αποκάλεσε ε, διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους να ξεκινήσουμε με το ΕΛΚ, τον Τόμας Μαν. Και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Κάρα. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς ε, την κυρία Βεντράουγκο από τον ΑΕΛΟ. Είπατε ότι δεν έχει περάσει ακόμα η κρίση και ότι οι πρώτες, ε, τα πρώτα θετικά μηνύματα δεν αρκούν. Γιατί πολλοί ακόμα ζουν στην φτώχεια και αυτό θα πρέπει να το αποτρέψουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα από τη Γερμανία. Θέλουμε μεσοκρατικών μέτρων να προωθήσουμε την σύντομη διάρκεια εργασίας για να ξεπεράσει ο κόσμος την κρίση και μετά όταν περάσει η κρίση να βρεθούν σε μια πιο πλεονεκτική θέση. Νομίζω ότι αυτό είναι βασικό θέμα και καλωσορίζω και αυτό το πακέτο εργασίας το κάναμε και στη χώρα μου αυτό. Υπήρχαν δηλαδή περιφερειακές ενώσεις για την εργασία, για να βρεθούν θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους. Ρωτώ το εξή λοιπόν. Από το Δεκέμβριο έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ενισχυθήκαμε στο ρόλο μας ως Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά ο χάρτης των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν έχει επικυρωθεί από τρεις χώρες. Ε, Θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί ένα δευτερεύον ζήτημα ή ένα πρωτεύον ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και σε επίπεδο ILO. Επόμενος ομιλητής, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Κάρας. Σας ευχαριστώ για τις αναλύσεις και για τις εκτιμήσεις σας. Στην Επιτροπή μας αντιμετωπίζουμε ασφαλώς το εξής πρόβλημα. Δεν θέλουμε να περιοριστούμε στην περιγραφή της κατάστασης. Θέλουμε να ε, δρομολογήσουμε και πολιτικές δράσεις. Και εδώ αντιμετωπίζουμε ένα όριο που έχει να κάνει με τις ε, διαφορές και τις ε, απαιτήσει που τίθενται στα κοινωνικά συστήματα. Τα κοινωνικά συστήματα φυσικά επαφείται στην ε, εθνική ερμοδιότητα. Έχουμε όμως και τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ιδιαίτερα σε θέματα των κοινωνικών θεμελιωδών δικαιωμάτων και της κοινωνικής ε, οικονομίας της αγοράς και της ε, απασχόλησης του ανταγωνισμού ως μέσο, όχι ως σκοπό, δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Εσείς, ε, ποιες απαιτήσεις μπορείτε να θέσετε έναντί μας. Πού θεωρείτε ότι θα πρέπει να περιοριστούμε σε συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία εντοπίζετε στην ανάλυση σας και πού από την πείρα σας θεωρείτε ότι οι εθνικές αρμοδιότητες θα πρέπει να εξευρωπαϊστούν προκειμένου να διασφαλιστεί αυτός ο ενιαίος, ο κοινός χαρακτήρας. Σε ποιον θα την ερώτηση, την ερώτηση κύριε Καράς. Θέλετε να αρχίσετε εσείς ε, κυρία Ουντράγκο. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση για τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, σίγουρα είναι σημαντική, αλλά ε, συνοδεύεται από παγκόσμιες ε, διατάξεις για την εργασία που έχουν προσπογραφεί από πολλές χώρες. Και η ΔΟΕ, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, προβλέπει ένα μηχανισμό για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής των ε, διεθνών κανόνων εργασίας. Και οι εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν κάθε ελευθερία να προσφύγουν στη ΔΟΕ και να ζητήσουν την γνωμοδότησή της για τις ε, υποτιθέμενες παραβιάσεις. Βέβαια η ΔΟΕ δεν ε, μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε μια χώρα, αλλά ακόμη και η ηθική πίεση που ασκείται με μια αρνητική έκθεση της ΔΟΕ είναι αρκετή για να διορθώσει πολλές ε, τασταλίες και παραβιάσεις των κανόνων εργασίας. Σας ευχαριστώ. Είναι θέμα περισσότερο νομικού πλαισίου πολιτικής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, γιατί οι συνθήκες προσδιορίζουν ότι τέτοιου είδου υπηρεσίε είναι οι δικές τους αρμοδιότητες. Πάντως, ε, το Κοινοβούλιο πρότεινε σε διάφορες κοινοβουλευτικές θητείες οι κοινέ ε, συμφωνίε των τοπικών και περιφερειακών αρχών, αν δεν ανταγωνίζονται τον ιδιωτικό φορέα και την ευρωπαϊκή αγορά, είναι δικό του θέμα. Αλλά δεν το δέχτηκε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν και κάποια ίσονο σημασία ζητήματα, τεχνικά μεν σημαντικά δε, που αφορά τι κρατικέ ενισχύσει για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Τώρα πάντω έχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο με το πρωτόκολλο για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στη συνθήκη της Λισαβόνας και εκεί ζητούμε διευκρίνηση του ισχύοντος πλαισίου και ένα υποστηρικτικό πλαίσιο πολιτικής για, την, ε, ε, για τη δημοκρατική αποκέντρωση στην Ευρώπη για να αποφευθούν κάποιες συγκεντρωτικές ή ε, κεντρομόλες τάσεις εξαιτία της κρίσης. Κύριε Σεράτκινς, μήπως θέλετε το λόγο. Όχι. Οπότε Συνεχίζουμε με τον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Γκέντς και μετά η Περβάνς Μπέρες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε καθηγητά Άτκινσον, είπατε ότι όλοι θεωρούμε ότι έχουμε πολλά στοιχεία για, το ΑΕΠ, αλλά, και την ανεργία, αλλά δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για τον πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο που έχει κρίση και το πώς επηρεάζει το βιωτικό επίπεδο του κόσμου. Έχουμε την αίσθηση ότι οι ανισότητες διευρύνονται και η συνοχή επίσης χαλαρώνει. Τα χάσματα ανοίγουν όλο και περισσότερο. Και πολλές φορές 20 με 40% των νέων μένουν άνεργοι. Βλέπουμε λοιπόν τον αντίκτυπο της κρίσης. Είπατε κύριε καθηγητά ότι έχουμε κάποια εργαλεία και πολιτικές για να βελτιώσουμε την κατάσταση και μερικοί οικονομικοί δείκτες φαίνεται να βελτιώνονται. Ερωτώ λοιπόν, ποια είναι η συμβουλή σας, τι προτάσεις μπορείτε να μας υποβάλλετε ώστε να βελτιώσουμε τις πολιτικές μας την κατάσταση αυτή. Η κυρία Μπερές. Η κυρία Γκέντς με πρόλαβε. Ακριβώς αυτή την ερώτηση θέλω να θέσω στον καθηγητή Άτκινσον. Πιστεύετε ότι είναι στα χέρια μας οι πολιτικές. Πολύ ευχαρίστω να κινητοποιηθούμε, αλλά τι ακριβώς πολιτικές, τι ακριβώς πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι πρέπει να αναλάβουμε. Μίλησατε για ένα διαζύγιο, για ένα ρήγμα που πραγματικά με τρομοκρατεί. Φαίνεται ότι δημιουργούνται κάποια διανετικά γκέτο μεταξύ το, του χρηματοπιστωτικού κόσμου και του λαού. Πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την αποκατάσταση των τραπεζικών περιθωρίων για να τα αξιοποιήσουμε και κοινωνικά. Σεράτκινσον. Πραγματικά κέρια ερωτήματα. τι πολιτικές ε, θα ήθελα. Σας μίλησα για το περσινό πακέτο Ομπάμα και σε ένα σεμινάριο ε, ε κάποιος ε, καθηγητής ζήτησε από έναν πρώην φοιτητή του που εργαζόταν στο Λευκό Οίκο και είπε στείλτε μου μια, ένα κατάλογο με τι θα επιθυμούσε. Το έκανε και περιλήφθηκε γιατί είπε ότι αποκλείεται να περιλαμβάνονταν όλα αυτά και όμως ζήτησε μια σειρά πρωτοβουλειών που τελικά περιλήφθηκαν και αυτά. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι λοιπόν. Σας είπα, θα μπορούσε να υπάρξει μια επέκταση του επιδόματος ανεργίας ή των κοινωνικών επιδομάτων. Νομίζω ότι και μόνο με αυτό θα αντιμετωπίσουμε πολλά ζητήματα θα πρέπει να διευρυθούν κάποια δικαιώματα. Βέβαια, η κοινή μακροοικονομία αυτό πρότεινε διαφοροποίηση των μεταφορών ανάλογα με το βάθος ε, της ύφεση. Επίσης μιλήσατε για τις επιπτώσεις τους νέους προηγουμένως. Ε, κάποιος ρώτησε και για τις εξουσίες ε, που υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά την πρόταση ενός εγγυημένου εισοδήματος για τα παιδιά. Ένα βασικό εισόδημα για τα παιδιά. Θα ήταν πραγματικά επένδυση για το μέλλον. Και πραγματικά ε, βοηθά μονογονικές οικογένειες ή χωρισμένους γονείς, γιατί αυτές είναι ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Μπορούμε να στήσουμε από τα κράτη-μέλη να προβλέψουν, να θεσπίσουν ένα τέτοιο ελάχιστο εισόδημα. Είχαμε διάφορες προτάσεις ε, για διατάξεις, για ελάχιστα εισοδήματα, αλλά αυτά είναι μέτρα που επαφίονται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Γιατί κάθε κράτο μπορεί να θετήσει διαφορετική λύση για το πώ θα δώσει σάρκα και οστά σε ένα τέτοιο ελάχιστο εισόδημα. Αν έχουμε όμω ένα ελάχιστο εισόδημα για τα παιδιά θα ήταν πολύ καλή απτή βοήθεια στις οικογένειες, αλλά και μήνυμα, σαφές μήνυμα της επιθυμίας της Ευρώπης να αναπτύξει την κοινωνική της διάσταση εν μέσω της κρίσης. Σε ό,τι αφορά το χρηματοπιστωτικό κλάδο και τις τράπεζες, δεν είμαι η δήμον για τις τράπεζες, αλλά πιστεύω ότι Πίσω από το θέμα αυτό κρύβεται ένα θεμελιώδες ερώτημα. Το πώς θα πρέπει να προσδιορίζουμε τις απολαβές, τις αποδοχές σε διάφορους τομείς ε, δραστηριοτήτων. Δεν είναι μόνο οι μισθή στις τράπεζες που ανησυχούν τον κόσμο. Μερικές φορές έχουμε χάσει τη, την αίσθηση τι σχέση πρέπει να έχουν ε, κάποιες υψηλόβαθμέ θέσει με τι αμοιβέ. Ποιε είναι οι αποδεκτές διαφορές σε τέτοιες θέσεις. Όχι μόνο για τους ε, εργαζόμενους στις τράπεζες, στο χρονομεταποστατικό κλάδο, αλλά και στους ακαδημαϊκούς κύκλους, ε, στα πανεπιστήμια. Και εκεί υπάρχουν ε, όλο και μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των χαμηλότερων και των υψηλότερων μισθών. Η πρόταση για την προοδευτική φορολογία εισοδήματο που έκανε ο κύριο Μόντι πραγματικά με βρίσκει σύμφωνο. σω είναι η ώρα να θεσπιστεί και ένα τέτοιο μέτρο. Να ρωτήσω τον κύριο Άτκινσον εξ ονόματο της ομάδας μου καταρχάς για την ε, πρόταση για την εξασφάλιση ενός ε, εισοδήματος ε, σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Ξέρω ότι στην χώρα μου γίνεται ε, μία ερώτηση, γίνεται ε, μία συζήτηση για την αύξηση του εισοδήματος και του επιδόματος για τα τέκνα. Το θέμα όμως είναι αυτό ωφελεί τελικά τα παιδιά ή μήπως ωφελεί ε, τον πατέρα τους που πίνει ενδεχομένως. αν θέλουμε να ωφελήσουμε τα παιδιά, αυτό είναι ένας στόχος που μας βρίσκει σύμφωνος στην Ευρώπη. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα να ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές, δηλαδή ε, παραδείγματα τα οποία επιτυχίας, που έχουν σταθεί με επιτυχία σε μια χώρα, να μην τα μεταφέρουμε στις άλλες χώρες. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όπως όλα τα θέματα των ε, αποδοχών και των ε, κερδών. Θα πρέπει να γίνει μια έρευνα για να δούμε πώς ε, ε, η αύξηση των επιδομάτων για τα παιδιά επηρεάζει την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Πολλές μελέτες γίνονται σχετικά. Πάντως ένα άλλο στοιχείο της συζήτησης αυτής, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ότι τα επιδόματα καταβάλλονται καταρχήν στις μητέρες, όχι στους πατεράδες και αυτό έχει μεγάλη συνέπεια. Μία από τις συνέπειες της, του προγράμματος Λισαβόνας ήταν η θέσπιση της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού στα κοινωνικά ζητήματα. Και εδώ μαθαίνουμε από τους ομολόγους μας. Και σε θέματα κοινωνικής προστασίας υπάρχει άμυλα και ο ένας μαθαίνει από τον άλλον. Βέβαια μερικές χώρες ε, έχουν καλύτερες επιδόσεις. Μερικές μείωσαν τελευταία πενταετία το ποσοστό φτώχειας τους. Ενώ άλλες δεν τα έχουν καταφέρει. Ίσως αυτές που έχουν μείνει πίσω θα πρέπει να παραδειγματιστούν από αυτές που είναι μπροστά. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι για το σημείο αυτό. Ένα από... Μία από τις συμβολές της Επιτροπής σας, τις συνεισφορές της Επιτροπής σας θα μπορούσε να είναι η αύξηση της δυνατότητας ανταλλαγής και αξιοποίησης των βέλτιστων πρακτικών δυνάμει του προγράμματος Λισαβόνας. Εκεί αναφέρονται κάπου οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, αλλά δεν αναμειγνύονται ενεργά. Ίσως αυτή η πιο ενεργός ανάμειξη για το μέλλον θα είναι πιο σημαντική. Επίσης, στις μελλοντικές συζητήσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα πρέπει να τεθούν όλα αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει το διαρθρωτικ... μόνο τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ανταλλαγής των πρακτικών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Πολύ χρήσιμο εργαλείο. Δύο, μιλητέ έχουμε ακόμα, την κυρία Φαρέρα και τον κύριο Καρφή. Σα ευχαριστώ. Ε, πείτε και σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας καλύτερα. Δύο ερωτήσεις έχω μία προς τον καθηγητή Άτκινσον και δεύτερη προς την κυρία Ουετράγο. Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι το ζήτημα που θέσατε είναι θεμελιώδες. Ποια είναι η γνώμη σας για το εξής. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις και έχουν πολύ διαφορετικές δυνατότητες και ικανότητες να παρατείνουν ε, τα μέτρα υποστήριξης για να αντέξουν στην κρίση. Ιδιαίτερα για τα κοινωνικά μέτρα μιλάω. Πιστεύετε, μήπως πιστεύετε ότι αυτές οι διαφορές θα επιταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν υπάρχουν ελάχιστες ευρωπαϊκές εσωτερικές πολιτικές για τα κοινωνικά ζητήματα. Κυρία Βεντράγκο, η Διεθνή Οργάνωση Εργασία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι όντω ένα ηθικό δεοντολογικό ζήτημα. Αλλά μήπω ήρθε η ώρα μέσα στην κρίση να έχουμε μια πιο άμεση σχέση μεταξύ τη Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου και των αρχών του ελεύθερου εμπορίου και των θεμελιωδών αρχών τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει ένα ανταγωνισμό επί τη ουσία και καταλήγουμε σε μία επιδείνωση των εργασιακών συνθήκων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλφιν. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω δύο ερωτήσεις προς τον καθηγητή Άτκινσον. Η πρώτη αφορά την φορολογική ε, ολοκλήρωση και βλέπουμε σε πολλά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το θέμα του συντονισμού. Μήπως χρειάζονται κάποια κοινωνικά κριτήρια και ορόσημα για τις κοινωνικές πολιτικές και τον κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης όταν μιλάμε επαναφορά σε ενοποιημένες, ολοκληρωμένες φορολογικές πολιτικές. Τι γίνεται με την, το είδος της οικονομίας που θα έχουμε στην ε, περίοδο μετά την κρίση. Θα έχουμε ανάκαμψη και επαναφορά στο προηγούμενο μοντέλο ή θα έχουμε μετάβαση σε ένα νέο είδος οικονομίας. Γιατί προσπαθούμε τη στρατηγική του 2020 να επικεντρώσουμε την οικονομία μας τις νέες τεχνολογίες, στην κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, την καινοτομία κτλ. Και τι γίνεται και με τις πολιτικές απασχόλησης. Όταν μιλούμε για πολιτικές απασχόλησης δεν πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την έλλειψη φορολογικών εργαλείων, να δούμε το είδος της απασχόλησης που επιδιώκουμε και τι πολιτικές απασχόλησης θα πρέπει να εφαρμόσουν οι χώρες για να τονώσουν την απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ σημαντικά και αυτά τα ερωτήματα. Για το τελευταίο σας σχόλιο, τις διαφορές στα κράτη-μέλη. Σίγουρα αυτές οι διαφορές είναι η αιτία πολλών ευρωπαϊκών θεμάτων και προβλημάτων. Όταν είπε για το ελάχιστο εισόδημα για τα παιδιά, ήταν ένα θέμα συναφέ με το βιωτικό επίπεδο σε κάθε χώρα. Αλλά βέβαια συστήγεται ένα ευρύτερο ζήτημα. Το ρόλο, τον ανακατανεμητικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη γίνεται τέτοια συζήτηση για τη σχέση μεταξύ του Κοινωνικού Ταμείου αφενός και του Ταμείου Περιφερειακής Συνοχής αφετέρου. Πέρυσι είχαμε μία μελέτη του κ. Πάρκερ για το ρόλο των Ταμείων συνοχή και πώς μπορούν να διευρυθούν και να εμπλουτιστούν με, ένα, με μία δέσμη κοινωνικών κριτηρίων. Πάντως και εγώ προ αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθούμε. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπε ερωτήσεις, ε, στη δεύτερη ερώτηση θα απαντούσα μονολεκτικά ναι, ότι χρειάζεται κοινωνική διάσταση στην φορολογική ενοποίηση. Τώρα τι μορφή θα πρέπει να πάρει αυτή. Αυτό προσπάθησα να πω και εγώ, ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση για τις συνέπειες και να προσθεθεί και ένα στοιχείο που παρέλειψε προηγουμένως, αλλά που διέπει όλη αυτή τη συζήτηση. Όταν μιλούμε για το κοινωνικό αντίκτυπο, εννοούμε αυτό το κάθετο αποτέλεσμα, διαφορά φτωχών και πλουσίων, αλλά υπάρχει και ένα αποτέλεσμα που διαπερνά τις γενναίες. Αυτό το αναφέρουμε και για τις κλιματικές αλλαγές. Πολλά θέματα που μας απασχολούν προϋποθέτουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν διαδοχικές γενιές. Αυτό ισχύει και για το θέμα της δημοσιονομικής ενοποίησης. Υπάρχει ένα φορτίο, αλλά πια γενιά θα το επομιστεί, η δική μου ή οι επερχόμενες. Και για τη συνδιάσκεψη που σας ανέφερα για το Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα πρέπει να προσθεθεί και μία διαγενειακή προοπτική. Και όταν μιλούμε για αύξηση της φορολογίας, θα πρέπει να δούμε πώς ε, οι επερχόμενες γιές θα αποφεληθούν. Ίσως η δική μου γενιά θα πρέπει να, καταβάλει ψηλότερη φορολογία για να χρηματοδοτηθεί εν μέρη και την πρόταση για το ελάχιστο εισόδημα παιδιών. Ε, και η δική μου γενιά θα πρέπει να πληρώσει ψηλότερους φόρους και ένα μωρό που είναι δύο ετών. Βέβαια, κάποιος από τις Βρετανικές αρχές στην επιστολή τώρα που είμαι 65 δεν χρειάζεται να, να πληρώνω την εθνική συνεισφορά. Δηλαδή, θα, χρειαστεί, θα μειωθεί η φορολογία. Με αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι σκανδαλώδες. Τώρα, για το είδο τη οικονομία. Ας μην ξεχνούμε ότι η σημερινή κατάσταση οφείλεται στις ε, αλλαγές της οικονομίας. Βρισκόμαστε σε μια πορεία αλλαγής. Και δεν πρόλαβα να αναφέρω όλα τα αποτελέσματα στην απασχόληση που οφείλονται στις αλλαγές στην αγορά εργασίας που έλεγαν χώρα την τελευταία δεκαετία. Γιατί ε, κινούμαστε σε μια πιο ευέλικτη αγορά εργασίας, χωρίς ταυτόχρονα να την ενισχύουμε με μια ασφαλή αλλαγή. Μιλούμε για flex security, αλλά περισσότερο δίνουμε έμφαση στο flex παρά στο security. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε από αυτή την προοπτική. Ευχαριστώ. Euh, Πολύ σύντομα για το πώς σχετίζονται ο ΠΟΕ με τον ε, δικό μας οργανισμό. Οι θεσμοί του Bretton Woods, η Παγκόσμια Τράπεζα και εμείς έχουν ορίσει μια πολύ θετική εξέλιξη εδώ και κάποιο διάστημα. Η κοινωνική ανάπτυξη και η ατζέντα της κοινωνικής ανάπτυξης ε, όλο και περισσότερο που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο προτεραιοτήτων αυτών των θεσμικών οργάνων. Υπάρχει ένα σύστημα διαρκών διαβουλεύσεων μεταξύ του ΠΟΕ, του, Παγκόσμιου, του, χρηματικού, του Νομισματικού Ταμείου, του δικού μας οργανισμού. Όλοι φροντίζουν να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και στην πράξη φροντίζουν να ευθυγραμμίζουν τις παρεμβάσεις τους. Έχουμε πολλά προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή για ζητήματα κοινωνική προστασία και συνεργαζόμαστε με την Παγκόσμια Τράπεζα, με το Παγκόσμιο με Νομισματικό Ταμείο εδώ και 1,5 χρόνια, χρόνο έχει ετοιμαστεί και κοινή έκθεση μεταξύ του δικού μας οργανισμού και του ΠΟΕ για τα θέματα του, τα εμπορικά, τα κοινωνικά και της κοινωνικής ανάπτυξης πιο συγκεκριμένα. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ότι με την ευκαιρία της κρίσης ή με αφορμή την κρίση, όλοι οι θεσμοί του ΟΗΕ προέβλεψαν εννέα πρωτοβουλίες που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Τομεί που έχουν πληγεί ιδιαίτερω από την κρίση, όπω η επιστημιστική ασφάλεια, η απασχόληση, το περιβάλλον και το καθεξής. Εκεί υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά όλοι αυτοί οι φορείς των διαφορετικών οργανισμών συνεργάζονται. Υπάρχει λοιπόν τεράστια πρόοδος από αυτή την άποψη. Για παράδειγμα, όταν ετοιμάζουμε εκθέσεις, όπως η έκθεση που προανέφερα, για τι τάσει τη απασχόληση φροντίζουμε να συζητούμε και με τον ΠΟΑ και με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και με την Παγκόσμια Τράπεζα, κάτι που προηγουμένω δεν γινόταν. Η κρίση λοιπόν ω προ αυτήν την έννοια μα ενίσχυσε τη συνεργασία μα. Από την άλλη πιστεύω ότι ω βουλευτέ και πρόσωποι των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε έναν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσετε. Και αυτό γιατί τα θεσμικά όργανα πολλέ φορέ καλούνται να συνεργαστούν. Τα κράτη-μέλη του το ζητούν. Και κάποιε φορέ ε, αυτό γίνεται και απαραίτητη προπόθεση. Από κάθε πλευρά λοιπόν έχουμε όλο και περισσότερε ευκαιρίε να ε, πετύχουμε σύγκληση απόψεων για πολλά ζητήματα, ιδίω ε, για τα θέματα τη ανάπτυξη. Σα ευχαριστώ και εξ ονόματο όλων μα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πανελίστε μα για τις εισηγήσεις τους. Μας δώσατε τροφή για σκέψη την οποία σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε στις μελλοντικέ μας εργασίες. Σας ευχαριστώ και να καλέσω το δεύτερο πάνελ. So, liebe Kollegen und Kolleginnen. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την δεύτερη, δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μας, της ακροασής μα ε, σε, ό,τι αφορά τις δημογραφικές ε, προκλήσεις και τα συστήματα συνταξιοδότησης. Έχουμε τρεις εξαιρετικούς εμπειρογνώμονες εδώ μαζί μας. Έχουμε την τιμή να τους έχουμε εδώ μαζί μα σήμερα. Καταρχάς, τον κύριο Edward Whitehouse, ο οποίος θα ξεκινήσει. Εργάζεται στον ΕΟΣΑ και είναι οικονομολόγος στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής, τον κύριο Βίτ Σάμεκ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και επικεφαλής ε, της νομικής υπηρεσίας στην Ομοσπονδία Συνδικάτων Τσεχίας Μοραβίας και τέλος έχουμε μαζί μας ε, εξ μου και την ε, κυρία γιατί θέλουμε πάντα να έχουμε και γυναίκες ε, πανελίστες, την κυρία Βιολέτα Τσουρέλ από τη Ρουμανία. Και οι τρεις έχουν διακριθεί ε, χάρη στις ε, δημοσιεύσεις, της, δημοσιεύσεις τους. Ανυπομονώ λοιπόν να ακούσω και τις εισηγήσεις τους και την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Το λόγο έχει ο κύριος Έντουαρντ Whitehouse. Αυτά λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ήθελα να αναπτύξω τα θέματα της έκθεσής μας συντάξεις με μια ματιά. Κάτι που ε, είναι έκταση 79 σελίδων, βέβαια, παρόλο που ονομάζεται με μια ματιά, έκδοση του ΩΣΑ. Και ήθελα να σταθώ κυρίω στι επιπτώσει τη κρίση εδώ ε, και έχουμε και τι 8 σελίδε τη ε, σύντομη έκταση που σα έχει υποβληθεί, για να τα διαβάσετε λίγο πιο σύντομα. Εδώ θα ξεκινήσουμε ένα παράθεμα από τους Financial Times κάτι που ανέφερε και ο Πρόεδρος σας το πρωί. Δηλαδή το θέμα του αν αυτή η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση θα μεταβληθεί σε κοινωνική κρίση ως προς τα ωφελήματα από, οποίο οποίο απολαύουν οι άνθρωποι κατά τη σύνταξή του, οι πολίτε κατά τη συνταξιοδότησή του. Το σημείο φετηρία τη ε, ήταν η χρηματοπροστατική κρίση, κάτι που φάνηκε να πλήττει τα συνταξιοδοτικά ταμεία και από το 2008. Αν δούμε του μέσου όρου, ε, φτάνουμε σε απώλειε του ύψου του 23%. Όμως, ε, οι απώλειε στι ΗΠΑ Πολιτείες ήταν κάπω υψηλότερε, ενώ ο σταθμισμένος μέσο όρο είναι 17%. Και φτάνουμε σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά σε χώρες όπως η Σλοβακία, η Τσεχία, η Γερμανία όπου έχουμε ιδιωτικά ταμεία συνταξιδότησης και που βασίζονται στην συλλογή των εισοδημάτων ε, από τι σύμφωνε φορέ των μελών του ε, αυτό φαίνεται ότι θα δώσει λιγότερε επιπτώσει για του ανθρώπου τη στιγμή τη αντικριτοδοτησής του. Κάποια στοιχεία τώρα αριθμητικά για την ανεργία και όπω είπε και ο κύριος Μόντι το πρωί για τι συντάξει: υπάρχει Υπάρχουν πολλά κενά πλέον στου ε, κρατικού προπολογισμού και σημαντικά ελλείμματα στι χώρε του ΩΣΑ. 8% αναμένεται για τα ερχόμενα τρία χρόνια. Και αυτό επηρεάζει σαφώς τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Πιέζει περισσότερο το, την πλευρά των ωφελημάτων βεβαίως, και για αυτό γιατί δεν έρχονται και τόσο συνεισφορές από τα μέλη των συντετοξιωτικών ταμείων. Η το βασικό μήνυμα από την ανάλυση μα και αυτό που θέλω να περάσω και όλα είναι ότι σε καμία χώρα το συνταξιωτικό σύστημα δεν θα παραμείνει αλόβητο από την ε, οικονομική κρίση. Όμω ε, ο αντίκτυπο διαφέρει γιατί η κάθε χώρα έχει το δικό τη συνταξιωτικό σύστημα και διαφέρει και βεβαίω για του πολίτε, του ίδιου του πολίτε μέσα σε κάθε μια χώρα. Η πρώτη μου παρατήρηση ε, έχει να κάνει με το ότι ενώ οι αποταμιεύσει για τα συντοξιστικά ταμεία είναι σημαντική πηγή για το εισόδημα κατά τη σύνταξη, οι ερευνητέ στις εβδομαδιαίες τους ε, εκδόσεις και σε ένα διάγραμμα που σα δείχνω εδώ στην οθόνη δείχνει το εισόδημα που θα προέλθει από τα ιδιωτικά συνταξιδοτικά ταμεία. Θα δείτε μια καμπύλη εδώ. Πιο ψηλά στον πίνακα έχουμε τις αγγλόφωνες χώρες ε, και την Ολλανδία, 40% των εισοδημάτων κατά τη σύνταξη από τέτοια ταμεία ιδιωτικά και μετά πολλά ευρωπαϊκά κράτη υπάρχουν στο κάτω μέρος του διαγράμματος και αυτό γιατί λόγου χάρη η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία είναι χώρες ε, που ξέφυγαν από τους οικονομολόγους ε, όταν εξέδωσαν αυτό το διάγραμμα, αλλά έχουν επιλέξει πολύ περισσότερο τα ιδιωτικά συνταξιδοτικά ταμεία πλέον και οι χώρες αυτές. Θα αλλάξει λοιπόν η εικόνα στο μέλλον. Η Ουγγαρία θα καλύψει το 1 τρίτο των συντάξεων από ιδιωτικά ταμεία στην ε, Τσεχία και την Σλοβακία παρόμοια ποσοστά. Εάν δούμε τώρα ένα δεύτερο σημείο πώς ε, επενδύονται οι αποταμιεύσεις των ανθρώπων σε επικίνδυνες, ε, όπως λέγονται, επενδύσεις, θα δούμε ότι το 2008, όπως φάνηκε και στην πρώτη διαφάνεια, υπάρχουν διαφορετικά κέρδη και θα δούμε πώς αυτό σχετίζεται με το χαρτοφυλάκιο των αξιογράφων των διαφορών χωρών. Στην Ιρλανδία υπάρχουν πολύ σοβαρές απώλειες λόγου χάρη, αυτό λόγω των ποσών που επενδύθηκαν ενώ στην άλλη άκρη του διαγράμματος, στην Σλοβακία και την Τσεχία υπάρχουν χαμηλότερες απώλειες λόγου χάρη, γιατί τα κυβερνητικά ομόλογα χρηματοδοτούν κυρίως τα συνδιοκτητικά ταμεία εκεί. Η εικόνα αυτή είναι όσο πιο επικαιροποιημένη γίνεται, αλλά τα στοιχεία που συλλέξαμε όπως ανέφεραν και κάποιοι από τους προλαλήσαντες, διέφεραν πολύ γιατί υπάρχουν χρονικά κενά στην περίοδο της κρίσης. Οι πληροφορίες κάποιες φορές είναι λίγο παλαιωμένες. Όμως υπάρχει ήδη μια ανάκαμψη, μέση ανάπτυξη 3%. Για τα συντοξιωτικά ταμεία το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι χώρε έχουν ήδη συλλέξει τα σχετικά δεδομένα, αλλά το δεύτερο εξάμεινο του 2009 υπήρχε περαιτέρω ανάκαμψη, ιδίω ε, στα ομόλογα και τα σχετικά αξιόγραφα. Σε ό,τι αφορά τι φορολογικέ πιέσει τώρα. Σε μερικέ χώρε ε, οι πιέσει είναι μεγαλύτερε, ιδίω όταν οι δημόσιε δαπάνε ήταν ήδη υψηλέ. Αυτό φαίνεται σε αυτό το διάγραμμα που βλέπετε μπροστά σα. Βλέπουμε ότι η Ιταλία και η Ισπανία έχουν 14% του εθνικού εισοδήματό του ε, να στηρίζεται στι συντάξει, στη Γαλλία το μισό περίπου, ενώ στο κάτω μέρο του διαγράμματο άλλα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιρλανδία 3,5%, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία στο 5% περίπου. Υπάρχουν μεγάλες φορολογικές πιέσεις, αλλά επειδή το ΑΕΠ μειώνεται και οι δαπάνες για τις συνταξιδοτήσεις δεν αυξάνονται παρομοίως, οι πιέσεις θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες στο μέλλον. Τώρα θα ήθελα να δούμε τα μακροχρόνια προβλήματα των συνταξιωτικών συστημάτων. Η οικονομική κρίση μα ε, έχει στρέψει περισσότερο στα βραχυπρόθεσμα προβλήματα, αλλά τα μακροχρόνια δεν θα εξαλειφθούν έτσι εύκολα. Γιατί μεταξύ άλλων έχουμε και τη γύρανση του πληθυσμού. Εδώ βλέπουμε την κυριότερη χώρα του ΩΣΑ στο διάγραμμα. Από το 2005 είναι η Ιαπωνία, την ακολουθούν από κοντά η Σουηδία και η Ιταλία. Και βλέπουμε εδώ να υπάρχει μια μεγάλη σύγκληση όλων των χωρών. Εδώ Τέσσερι άνθρωποι σήμερα εργάζονται για έναν συνταξιούχο γύρω στα 30 του, ενώ πολύ σύντομα το 2030 θα έχουμε φτάσει σε τρει για τον ίδιο συνταξιούχο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγάλο φορολογικό κόστο από την χρηματικοπιστωτική και οικονομική κρίση με την γύρανση των εργαζομένων. Ε, με του υπολογισμού μου βλέπουμε, είδα ότι το μέσο όρο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου όλο ένα και μειώνεται και το κόστο θα δεκαπλασιαστεί το φορολογικό κόστος, θα δεκαπλασιαστεί από τις συντάξεις, ε, για τι συντάξει μάλλον εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Άρα οι άνθρωποι τη ηλικία μου φαίνεται ότι θα επηρεαστούν από τα συμπεράσματα της πολιτικής μας. Οι χώρες που ε, έχουν δώσει σκληρούς πολιτικούς αγώνες στο παρελθόν και έχουν πετύχει συνταξιδοτικέ μεταρρυθμίσει μπορεί να τα καταφέρουν, αλλά μπορεί και να χρειαστεί να μεταβάλουν τις μεταρρυθμίσεις τους αυτές. Οι συνταξιούχοι που θα χρησιμοποιούν τα ωφελήματα της σύνταξης, αναπηρίας και άλλο επιδόματα ανεργίας, όλα αυτή, ο, ο, ο αριθμός τους θα μειωθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και σε σχέση με τη δεκαετία του 80 που υπήρχε παρόμοια ύφεση. Είχα, είχαν χρειαστεί δύο δεκαετίες εδώ για να αυξηθούν τα ωφελήματα αυτά και να στηριχθεί η αγορά εργασίας, αλλά η οικονομική κρίση επηρεάζει και τις επενδύσεις στα συντοξιδικά ταμεία. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι στα συστήματά μας που αντιμετωπίζουν τα άτομα μεμονωμένα αλλά και το σύστημα συνολικά. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί διαφοροποίηση για τι διατάξει των συνταξιωτικών ε, συστημάτων ανάλογα με του διαφορετικού κινδύνου που αντιμετωπίζονται. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Σάμεκ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είμαι σε πλεανεκτική θέση γιατί ο προηγούμενος ομιλητής ε, παρουσίασε πολλές από τις πληροφορίες τις οποίες θα ήθελα να σας δώσω και εγώ. Γι' αυτό θα περιοριστώ στο κοινωνικό αντίκτυπο των συνταξιοδοτήσεων και την ε, επιρροή της κρίσης στις συνταξιοδοτήσεις. Βλέπουμε τις πηγές εισοδήματος στις μεγάλες ηλικίε και υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Οι χώρες της ε, Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης ε, έχουν ε, έχουν διαφορετικές πηγές σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους. Άρα οι μεταρρυθμίσεις που αναφέρει ο συνάδελφος αναγκάζουν τις χώρες αυτές σε πολλές περιπτώσεις να μεταφέρουν χρήματα από δημόσια συστήματα σε ιδιωτικά. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο στήλες ε, σε κόκκινο χρώμα. Βλέπουμε το μέσο εισόδημα, μισθό και στην τσεχική δημοκρατία Κοιτάξτε. Από το 1,1 στο 1,5. Πάνω από το 1 πέμπτο του πληθυσμού στην Τσεχία έχουν καλούς μισθούς. Γι' αυτό λοιπόν ε, ε, μπορεί να μην γίνει τέτοια μεταφορά από τα δημόσια συστήματα στα ιδιωτικά συστήματα. Η γύρανση είναι ένας προβλεπόμενος κίνδυνος, ο οποίος είναι συγκρίσιμος με την κρίση, αλλά είναι πιο προβλέψιμος από την ε, χρηματοοικονομική κρίση. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε ότι θα είναι πιο εύκολο να επιλύσουμε τα προβλήματα των δημόσιων συστημάτων σε σχέση με τα προβλήματα των ε, ιδιωτικών συστημάτων. Υπήρξε αλλαγή, για παράδειγμα, των παραμέτρων από 63-65 έτη στο όριο τοξιδιώτησης. Και στην μπλε γραμμή βλέπετε το θετικό αντίκτυπο για την ε, οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος μας. Ένα παράδειγμα οικονομικής κρίσης και του αντίκτυπού της είναι το εξής. Βλέπετε την κόκκινη γραμμή η οποία αποτελεί την προοπτική του, του συστήματος αξιοδότησης πριν, αλλάξει, πριν αλλάξουν οι παράμετροι. Πριν λάβουμε υπόψη, δηλαδή, τον αντίκτυπο της κρίσης. Λέμε λοιπόν ότι δεν ε, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Μπορούμε να αλλάξουμε τα ιδιωτικά, τα δημόσια συστήματα σε ό,τι και τα κοινωνικά δικαιώματα που συνεπάγονται τα συστήματα αυτά. Είπε ο συνάδελφο ότι υπάρχει το πρόβλημα των συνταξιωτικών ταμείων, γιατί ενδεχομένω να είναι πολύ διαφορετικέ οι συνθήκε. Και ίσως ε, να μην αναμενόταν να κινηθούν σε τόσο θετική κατάσταση, σε τόσο θετική κατεύθυνση τα ιδιωτικά ταμεία. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρουσίαση έγινε πέρσι από τον Μάικλ Σισόν στην Πρατισλάβα για τον αντίκτυπο της κρίσης στα διάφορα συνταξιδευτικά συστήματα. Το μήνυμα του κυρίου Σισόν ήταν πολύ παρόμοιο με το δικό μου μήνυμα. καταδεικνύεται σαφέστατα ο αντίκτυπος στο μεμονωμένο συνταξιοδοτούμενο. Συγκρίνοντας τις απώλειες που σημειώθηκαν, που είναι πάρα πολύ υψηλές και συνεπάγονται την καταστροφή των επενδυτών. Γιατί αν για παράδειγμα είναι κανείς 58-59 ετών και τον χτυπήσει η κρίση. Το αποτέλεσμα το περιέγραψε ο ΣΑ. Είναι τεράστιο και καταστροφικό το αποτέλεσμα. Χάνει κανείς το χρήματά του, χάνει τη μελλοντική του σύνταξη. Και ο κύριος Σισόν παρέθεσε πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για την απόκριση την πολιτική, πολύ διαφορετική σε διάφορα τμήματα του κόσμου, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία, και σε πολλές άλλες χώρες, σε κάποια συστήματα υπάρχει ε, εκ νέου κρατικοποίηση των συνταγματικών, των συνταξιδευτικών ε, συστημάτων Ποια, ποιο είναι το μέλλον τώρα των συνταξιευετικών ε, συστημάτων σε ό,τι αφορά την ένωσή μας. Υπάρχουν δύο σενάρια. Η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο άσκησαν ε, πιέσεις για να μειωθούν οι εισφορές και να δίνεται μικρό τμήμα των χρημάτων αυτών, δηλαδή να αντικατασταθούν τα συστήματα αυτά σε περιορισμένο βαθμό. Να προσθεθούν λοιπόν χρήματα στο σύστημα. Πέρσι αναφέρθηκαν πολλά στοιχεία για την ανανέωση του συστημάτων Pay As You Go. Για να υπάρχουν βιώσιμες ε, συνταξιοδοτήσεις. Τα... Το δεξί σενάριο συνεπάγεται ισχυρό σύστημα Pay As You Go. Για παράδειγμα, λοιπόν, υπάρχει εξή κατάσταση στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ποιος μπορεί να συνδράμει τι στα συστήματα. Προς το παρόν έχουμε 0% σε ό,τι αφορά τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις και μετά ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν κάποιες εισφορές ε, στα συστήματα για να προσθέσουμε συμπληρώματα στα συστήματα pay η σλοβάκικη περίπτωση όπου υπήρχε opting out τα ελλείμματα το οποίο προκαλούνται από τέτοιες καταστάσεις είναι υπερβολικά υψηλά και δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον της Σλοβακίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, αλλά είναι τεράστιος ο κίνδυνος που υπάρχει. Και γι' αυτό και είμαστε κατά τέτοιων μεταρρυθμίσεων. Το καλύτερο σενάριο και το μοναδικό, αν θέλετε, για τη μεταρρύθμιση της, ε, των συνταξιτικών συστημάτων είναι η μετανάστευση και το να κάνει ο κόσμος πολύ πιο πολλά παιδιά. Yeah. Σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου χαρά που έχω την ευκαιρία να αναπτύξω κάποια από τα συγκεκριμένα ζητήματα που ε, αφορούν τα συνταξιωτικά ταμεία των κεντρικών ε, ευρωπαϊκών κρατών, μάλλον των κρατών της κεντρικής Ευρώπης. Κάποιες από τις πτυχές που θα ήθελα να αναπτύξω στην παρουσίασή μου ε, έχουν ήδη αναφερθεί από τους προαλήσαντες, οπότε δεν θα τα επαναλάβω. Απλώς θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στην πολιτική διάσταση, κυρίως για το πώς μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη προσέγγιση και σε σχέση με τη γέννηση του πληθυσμού και τις δημοκρατικέ μεταβολές. Είναι πολύ σαφές ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης μειώνεται, συρρυκνώνεται. Ο, το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται, η γύρανση του πληθυσμού είναι κάτι που και προηγουμένως το αναφέρατε, επανειλημμένος. Και για την γύρανση του πληθυσμού βλέπουμε ότι και οι περισσότερες χώρες ε, θα πληγούν λόγω του φαινομένου αυτού. Ίσως η Ευρώπη μετά την Ιαπωνία είναι η γυρεότερη περιοχή του κόσμου και μάλιστα γυράσκει με πολύ γοργούς ρυθμούς. Τώρα, για τη γύρανση πρόσφατα διάβασα σε ένα πολύ ενδιαφέρον, ένα πολύ ενδιαφέρον του κ. Τζανίνη από την Γενέβη, όπου γίνεται λόγος για Ίσως ανανέωση ή νέα γενιά ανθρώπων, ιδίως γιατί συνταξιούχοι μετά τη συνταξιοδοτησία τους μπορεί να έχουν και πολύ έντονη ζωή. 70 έως 80 οι 70χρονοι και 80χρονοι σήμερα, ε, σε σχέση με ανθρώπους που στην αρχή του αιώνα ήταν 20 χρόνια νεότεροι τους, ε, έχουν πλέον πολύ πιο έντονη ζωή. Πάντως, η γύρανση του πληθυσμού μπορεί να εξεταστεί και σε σχέση με τα φαινόμενα μετανάστευσης και πώς μπορεί να μετριαστούν οι τάσεις γύρανσης μέσω την έλευση μεταναστών. Εδώ να παρουσιάσω την περίπτωση της Ρουμανίας, επειδή είμαι Ρουμάνα Η αναλογία 4 προς 1 της Ευρώπης αναμένεται το 2060 να έχει φτάσει στο μισό, στο 2 προς 1. Στην περίπτωση της χώρας μου, τα ποσοστά αυτά θα μειωθούν πάρα πολύ. Ακόμη λοιπόν και αν οι αριθμοί είναι πολύ ανησυχητικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήδη το 2009 Είχαμε αναλογία 1% για το ποσοστό εργαζομένων που εργάζονται ένα συνταξιούχο. Και το 2015 θα είναι 0,4 προς 1. Βλέπετε ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος πολιτικός ό,τι αφορά την προσέγγιση των, των συντάξεων. Σίγουρα υπάρχουν και τεράστιες διαφορές μεταξύ των παλιών και των νέων ευρωπαϊκών χωρών σε ό,τι αφορά τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και αυτό ε, δημιουργεί τεράστιες πιέσεις στις επιχειρήσεις, στους κράτους, στα κράτη, στους κρατικούς προϋπολογισμούς αλλά και στους ιδιώτες. Τώρα, αν εξετάσουμε τι ε, κεντροευρωπαϊκές χώρες, ε, τα συνταξιδοτικά ταμεία, καταρχήν οι περισσότερες έχουν ιδιωτικά συστήματα και κρατικά συστήματα στα εξοδοτικά. Εκεί οι αποδόσεις ήταν αρνητικές το 2008 όπως παντού άλλωστε, οπότε σε σύγκριση με τις χώρες του ΩΣΑ, το 23, 23, λίγο, ε, μείον 23% ε, αν εξαιρέσουμε τις Ηνωμένες που είναι μείον 17%. Τώρα, σε σχέση με το παγκόσμιο επίπεδο, μείον 18% για το 2010 και στη, στην κεντρική Ευρώπη ο μέσος όρος ήταν καλύτερος για τα συνταξιδοτικά ταμεία, μείον 13%. Ε, το 2009 βλέπετε ότι σχεδόν όλα είναι πράσινα, άνω του μηδενός δηλαδή. Είχαμε θετικές επιστροφές για το 2009 σε όλες τις χώρες. Και αν κοιτάξουμε και την αξία των ε, στοιχείων του ενεργητικού, των καθαρών, βλέπω ότι στο τέλος κάθε περίοδου είχαμε αύξηση μάλιστα το 2009. Αυτό οφείλεται στις συνεισφορές αλλά και στις επιστροφές τα κέρδη των επενδύσεων. Βέβαια, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο. Πολλές αρνητικές δράσεις έληφθησαν από τις κυβερνήσεις σε πολλές από τις κεντροευρωπαϊκές χώρες Έχω και ένα παράρτημα στην έκθεσή μου με λεπτομεριακές περιγραφές για κάθε χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, αν σας ενδιαφέρει. Και αυτό συνέβη άσχετα με τις ε, προηγούμενες επιδόσεις των συνταξιδοτικών ταμείων. Είχαμε μειώσει τις συνεισφορές και επίσης ανώτατα όρια για τους παρόχους συντάξεων. Βέβαια και οι πολιτικές αποφάσεις μερικές φορές ε, επηρέασαν τις ε, αποδόσεις των συντάξεων. Τι κίνδυνοι υπάρχουν, όπως φάνηκε και από την κρίση, ο πιο εμφανής κίνδυνος για τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα, γενικώ για τα συνταξιοδοτικά συστήματα, κρατικά και ιδιωτικά, ιδιωτικά είναι ο πολιτικός κίνδυνος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόσκομα για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των συνταξιδοτικών συστημάτων στην Κεντρική Ευρώπη. Ο πολιτικός κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος από το επενδυτικό κίνδυνο, από τα προβλήματα της ανεργίας, αλλά και τις άλλες κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Νωρίτερα συζητήσαμε και τη διαφοροποίηση του κινδύνου και την μη διακριτική μεταχείριση των συντάξεων. Δεν θα επιμείνω σε αυτό, πάντως είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε αυτό το εξάμεινο που η πάταξη των διακρίσεων αποτελεί και προτεραιότητα της ε, Ισπανικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα η διαφοροποίηση είναι σημαντική ως προς την έκθεση στον κίνδυνο. Και πολλοί είναι οι κανονισμοί αλλά και οι οδηγίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν ε, και τις ασφάλειες ζωής. Αλλά, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να δούμε την ασφάλεια ζωής σε κάθε χώρα χωριστά εξαιτία των διαφορών. Αν εξετάσουμε τον αντίκτυπο της κρίσης στις επιχειρήσεις και τους πελάτες, η μεγαλύτερη επίπτωση είναι η μείωση των συνεισφορών εξαιτία ε, τη χαμηλή απασχολησιμότητα και όχι επιστροφέ ε, ή τα κέρδη των συνταξιδοτικών ταμείων, που επαναλαμβάνω δεν ήταν τόσο λιγότερα από το 2008. Υπάρχει επίσης μια αναδιαμόρφωση του τοπίου του ανταγωνισμού. Οι πελάτες έχουν χάσει χρήματα, δεν ξέρουν σε ποιον να επιρρύψουν την ευθύνη. Πάντως, σίγουρα δεν έγινε προσπάθεια σωστής ενημέρωσης, διαπαιδαγώγησης και από την πλευρά των κυβερνήσεων, αλλά και από την πλευρά των οργανώσεων προστασίας του καταναλωτή, για να είναι πιο ενημερωμένοι, πιο καταρτισμένοι, πιο κατατοπισμένοι οι επενδυτές για την πορεία των επενδύσεων, για να ξέρουν ε, τι κινδύνους αναλαμβάνουν. Δεν έχω αρκετό χρόνο για να εξετάσω όλα τα θέματα και τις μελλοντικές προοπτικές. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να πω ότι στην κεντρική Ευρώπη τα συνταξιδοτικά ταμεία μάλλον βγήκαμε το κεφάλι ψηλά από την κρίση σε σχέση με άλλες περιοχές ή χώρες. Βέβαια υπάρχει πολύ απτός δημογραφικός κίνδυνος και όλοι οι δείκτες και τα στοιχεία που εξετάστηκαν νωρίτερα οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα ότι χρειάζονται οπωσδήποτε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να βοηθήσουμε τον γυράσκοντα πληθυσμό να κάνει τη μετάβαση, αλλά και μακροπρόθεσμα χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές. Επίσης το εργατικό δυναμικό θα συρρυκνωθεί, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ο οικονομικός παράγοντας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μόνο υπέρ τη μεταρρύθμιση των εξαιρετικών ταμείων, αλλά και το Διεθνέ Ομοσπονδιακό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα και όσα. Οι κρατικέ συντάξει δεν είναι βιώσιμο μέτρο εξαιτία των λόγων που αναφέραμε. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε σημαντικέ μεταρρυθμίσεις και σε καμία περίπτωση υπανοχώρηση τη της κατάστασης των περσινών ετών. Η ανεργία φυσικά είχε σημαντικό αντίκτυπο, αλλά και ο δημοσιονομικός αντίκτυπος διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα και με την επίδοξη του συνταξιδοτικού ταμείου, αλλά και με τη διάρθρωση του συνταξιδοτικού συστήματος σε κάθε χώρα. Και κάθε, κάτι που κατά τη γνώμη είναι πολύ σημαντικό και προφανέστατο, και θα ήθελα να το επαναλάβω και να το διατρανώσω, είναι η... μερικές φορές η βραχυπρόθεσμη προοπτική των κυβερνήσεων. Είναι μέσα μερικέ φορέ οι κυβερνήσει ό,τι αφορά τι ταξιδοτικέ μεταρρυθμίσει. Γιατί τέτοιε μεταρρυθμίσει απαιτούν ε, μεγάλη οικονομική προσπάθεια και υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί. Βέβαια, κάθε πολιτικό θα πρέπει να είναι διορατικό και να βλέπει πιο μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι προ όφελο και τη χώρα αλλά και του κόσμου. Αν ε, είναι πολύ κοντόφθαλμε οι βραχυπρόθεσμε οι αποφάσει ε, και δεν ξεπερνούν μία πενταετία, δεν είναι βιώσιμες δεν είναι καλές. Να μην πω τίποτα χειρότερο. Ο ρόλος τέτοιο βραχυπρόθεσμα και κοντόφθελων μέτρων είναι κατάλληλος. Ο πολιτικός θα βλέπει να είναι πιο διορατικός, να βλέπει πιο μακριά. Ο πολιτικός κίνδυνος λοιπόν είναι σαφής. Για να αναφέρω ακροθυγώ και μερικέ λύσει. Ανάγκη βιώσιμων μεταρρυθμίσεων που θα εστιάζονται σε μακροπρόθεσμη προοπτική. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητε. και να δούμε πώς θα προσαρμοστεί ο γυράσκο πληθυσμό και να υποστηριχθεί ε, ο κόσμος, να μπορέσει να πραγματοποιήσει την μετάβαση εισαγωγή και στήριξη επικουρικών στεξιδοτικών συστημάτων, κατάλληλες φορολογικές προσαρμογές και ενημερωτικά προγράμματα, προγράμματα σωστής διαπαιδαγώγησης και κατατοπισμού των πολιτών. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, των εποπτικών αρχών και των νομοθετών, καθώς και όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο διάλογο. Και τέλος, ευρωπαϊκό επίπεδο, ίσως θα ήταν σκόπιμο να υιοθετήσουμε μια πανευρωπαϊκή θεώρηση των συντάξεων. Κάτι που θα δώσει ενάβσματα και σε μεγαλύτερη κινητικότητα. I'm happy to answer. Ε, είμαι στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσω σε απορίες σας. Έχω και ένα παράρτημα πολύ λεπτομεριακό που δείχνουν ότι η κατεύθυνση και των κεντροευρωπαϊκών χωρών δεν είναι και πολύ καλή γιατί προσπαθούν να επανέλθουν σε κρατικές συντάξεις ή προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες α, επιστροφές ή κέρδη των συντάξεων για να επιλύσουν βραχυπρόθεσμα κάποια προβλήματα. Αυτός είναι λάθος δρόμος. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι θα πρέπει να φύγει σε λίγο η κυρία Περές, η οποία είναι και η συγγήτρια, γι' αυτό θα της δώσω κατευθείαν το λόγο και μετά θα ακούσουμε τους ε, υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ θερμά και το πάνελ. Ήταν πολύ χρήσιμες ε, οι ομιλίες αυτές και πολύ διαφωτιστικές. Κύριε Σιουρέλ, είμαστε μια ομάδα σοσιαλιστική. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν αυτά τα πράγματα και δεν σκεφτόμαστε μόνο το κοντόφθαλμο και τις επόμενες εκλογές και το να επανακλαγούμε. Σίγουρα ήταν πολύ βραχυπρόθεσμες οι λύσεις που ελήφθησαν όχι μόνο από κυβερνήσεις αλλά και από χρηματοπιστωτικούς παράγοντες και αυτό οδήγησε την οικονομία μας στην κατάσταση που έφτασε σήμερα. Και όχι μόνο την ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια. Ακριβώς αυτός ο κοντόφθελμος και βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας. Κύριε White Whitehouse, βλέποντας τον πίνακα αυτό και συγκρίνοντάς τον με το δικό σας, διαπιστώνω ότι έχουμε να λύσουμε μία εξίσωση ανεπίλητη γιατί το δημόσιο χρέος ε, περιπλέκει τα συστήματα, τα συνταξιοδοτικά, αλλά και η σύνταξη με την κεφαλοποίηση δεν είναι κατάλληλη λύση. Ε, Δυστυχώ ο συνάδελφος Ρίχαρτ Φάλμπρ έφυγε. Ε, έχω μια ερώτηση όμως δική του να σας διαβιβάσω. Θεωρείτε ότι η διαχείριση των συνταξιοδοτικών ταμείων με κερδοσκοπικό τρόπο συνέβαλε στην κρίση που ζούμε σήμερα. Και δεύτερον, όπως μας είπε και ο κύριος Σάμεκ, θα πρέπει να ενισχύσουμε το δεύτερο και τρίτο πυλώνα των συνταξιδοτικών συστημάτων, αλλά μόνο με κάποιους μηχανισμούς διακυβέρνησης και κρατικού προσδιορισμού των μακροπρόθεσμων επενδύσεων που θα είναι κρίσιμες. στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου ήταν ε, αδύνατον να επισέλθω σε πιο πολλές λεπτομέρειες ε, για το ερώτημα αυτό και προφανώς ε, δεν μπορούν να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις βάσει των αποδόσεων ενός έτους για τα σταξιδικά συστήματα. Κοιτώντας μακροπρόθεσμα, οι αξιογράφα είχαν απόδοση περίπου 7% ανά έτος, επειδή μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό μας ενδιαφέρει και σαφώς υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει κόσμος ο, οποίος λίγο πριν τη συνταξιοδότηση δεν μπορεί ούτε να δουλέψει παραπάνω ούτε μπορεί να κάνει αποταμίευση για να αντισταθμίσει τις απώλειες αυτές. Στην παρούσα φάση προτείνουμε στις πιο πολλές χώρες να έχουμε μία ενιαία ε, επενδυτική στρατηγική. Και άρα ο κόσμος που ετοιμάζεται να βγει ε, στη σύνταξη έχει μεγάλο τμήμα των επενδύσεών του στην ε, κεφαλαγορά. Στο χρηματιστήριο. Και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιος αυτόματος μηχανισμός προκειμένου να μεταφερθούν σε πιο λιγότερο επικίνδυνες επενδύσεις τα χρήματα και αποταμιεύσεις του κόσμου που ετοιμάζεται να βγει στη σύνταξη. Θα πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν διαφορετικά, διαφορετικές επενδύσεις με διαφορετικό κίνδυνο και αυτόματα να μεταφέρεται ο κόσμος όσο πλησιάζει τη σύνταξη σε λιγότερο ε, επισφαλείς επενδύσεις. Βλέπουμε ότι έχουμε διάφορα συστήματα συνταξιοδότησης και γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να βάζει κανείς όλα τα κεράσια σε ένα καλάθι, αλλά να κάνει κατανομή του κινδύνου και των επενδύσεων του. Τα ιδιωτικά συστήματα που επικρατούν σε πολλές χώρες σήμερα πρέπει να επανεξεταστούν. Μία ερώτηση από το ΕΛΚ. Υπάρχει κανείς που θέλει να θέσει ερώτημα από το ΕΛΚ. Ο κύριος ε, Κάρας. Ναι, υπάρχει μία ενιαία γραμμή και για τα κοινωνικά συστήματα και για τα συστήματα τα συνταξιβατικά. Καταρχάς, αρμόδια είναι, στο πρώτο πυλώνα, αρμόδια τα κράτη-μέλη. Δεν ε, ε, ανάλογη συμμετοχή του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα σε ό,τι αφορά τη συνταξιδότηση. Και γι' αυτό είναι και άνηση η σχέση μεταξύ των κρατικών συστημάτων που είναι όλα υπερχρεωμένα. Και έχουμε και τα ιδιωτικά συστήματα, τα οποία έχουν υποστεί τις πιο μεγάλες απώλειες, γιατί υπάρχει περιορισμένη ευθύνη. Και αυτό αποτελεί συνέπεια της κρίσης. Αλλά πέρα από την κρίση υπάρχει και η δημογραφική εξέλιξη, την οποία θα πρέπει να επιλύσουμε. Τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει αφενός να κοιτάξουμε τι, πώς τα συστήματα μας θα, θα εξασφαλίσουν τη συνταξιδοτική ασφάλεια βάσει των δημογραφικών αλλαγών, αφενός λοιπόν, και στο, στη δεύτερη φάση θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να ενισχύσουμε κατά τη μεταρρύθμιση αυτή, προκειμένου να εξάλθουμε και από την κρίση, γιατί η κρίση ουσιαστικά όξινε το πρόβλημα της ε, δημογραφικής εξέλιξης. Και τώρα λοιπόν το μεγάλο ερώτημα που ανακύπτει είναι ότι δεν έχουμε το σύστημα των τριών πυλώνων σε ένα κράτος μέλος. Και το θέμα του αυτοματισμού. Για παράδειγμα, στο δεύτερο πυλώνα, το οποίο αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ότι στο τρίτο πυλώνα. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνουμε προκειμένου τα συστήματα να είναι συγκρίσιμα στα κράτη-μέλη, Πού μπορούμε να ακολουθήσουμε ευρωπαϊκή προσέγγιση και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μην τα απαλλάξουμε για την ευθύνη τους ε, στον πρώτο πυλώνα και μπορούμε να ενισχύσουμε πιο εύκολα τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα από τον πρώτο. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής προκειμένου να πετύχουμε να πραγματοποιήσουμε αυτά που προτείνεται Και απευθύνω την ερώτηση αυτή και στους δύο μιλητές. Uh, Κοιτάξτε, κάναμε μια πρόταση για πανευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις συντάξει στον τρίτο πυλώνα. Προσπαθήσαμε να δούμε και το δεύτερο πυλώνα και είχα στείλει σχετικά την πρόταση και ήταν εδώ στο τραπέζι. Είναι μάλλον να σας ενδιαφέρει. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που εντοπίσαμε για να, κάνουμε, για να βρούμε κάτι το οποίο να εφαρμόζεται γρήγορα. Ήταν οι διαφορές οι φορολογικές, κάτι που συζητήθηκε σήμερα. Όμως αν υπάρχει πολιτική βούληση, ήταν εκεί και η κυρία Μπερέζ όταν ξεκίνησε η έρευνα, το τέλος του 2007. Αν υπάρχει λοιπόν πολιτική βούληση όπως έλεγα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στον τρίτο πυλώνα ε, θελοντική αποταμίευση. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Και είναι και θέμα κινητικότητας εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αν αυξηθεί κινητικότητα, πώς θα λειτουργήσει η φορολόγηση για το δεύτερο πυλώνα. Αν δούμε αντικειμενικά τα εμπόδια που υπάρχουν, ο στόχος είναι πολύ μακροπρόθεσμος. Έτσι πρέπει να τον δούμε. Ο ορισμός των πυλώνων είναι διαφορετικός. Αν δείτε τις παλιές ευρωπαϊκές χώρες. Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα θέματα απασχόλησης. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δεύτερος πυλώνας, ε, περιέχει υποχρεωτικά μέτρα όσον αφορά τις αποταμιεύσεις στο πολωνικό μοντέλο και παρόμοια σε άλλες χώρες, Σλοβακία, Ρουμανία. Τρίτος πυλώνας είναι οι ε, θελοντικές ε, αποταμιεύσεις. Διαφέρει σε χώρες. Καμιά φορά είναι αποκλειστικά τομικές αποταμιεύσεις, αλλού συνεισβάλλουν και οι εταιρείε. Σε χώρες όπως η Ουγγαρία θέλουν να οι διευκολύνσει όσον αφορά τι εθελοντικέ ε, εισφορέ θέλουν να καταργηθούν. Από κάτι θα επηρεάσει τι οικονομίε τελικά, τι ατομικέ. Μόνο για τον τρίτο πυλώνα κάτι μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Εγώ αυτό πιστεύω για το δεύτερο πυλώνα μια ευθυγράμμιση των συστημάτων ίσως να συμβεί στη γενιά των παιδιών μας, όχι στη δική μας εποχή. Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η απόψή μου. Να προσθέσω, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον πρώτο πυλώνα όσον αφορά τα συνταξιωτικά συστήματα των κρατών μελών. Έριξα μια ματιά στο Ηνωμένο Βασίλειο Ορισμό αντικατάσταση του πρώτο πυλώνα είναι περίπου 30% στην Ιρλανδία, 35%, Σουηδία 38%. Και αν τα συγκρίνεται με την Αυστρία και την Ισπανία, ε, υπάρχει τεράστια διαφορά. Υπάρχει μεγάλο φάσμα μέτρων του πρώτου πυλώνα και σε χώρους όπως η Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο που πάντα υπάρχουν προγράμματα, υπήρχαν προγράμματα μικρά στον πρώτο πυλώνα, πάντα υπήρχε η παράδοση το εργατικό δυναμικό στην πλειοψηφία του να καλύπτεται από ιδιωτικά συνταξιωτικά ταμεία. Ένα από τα βασικά εμπόδια για πανευρωπαϊκή λύση, για συνταξιωτικό μοντέλο πανευρωπαϊκό, είναι ότι παρέχονται διαφορετικό τρόπο οι συντάξει στι διάφορε χώρε. Στην Ολλανδία, 95% ε, είναι τύπου εισφορών. Η Ιρλανδία και η Βρετανία ήταν του καθορισμένης μάλλον ευεργητημάτων και πάνε προς καθορισμένες εισφορές. Οπότε επικίνουν τα συστήματα. Οι εταιρείε που δουλεύουν σε διάφορα κράτη-μέλη θα διευκολυνθούν αν κινούνται στα πλαίσια ενός συνταξιωτικού συστήματος και η Ευρωπαϊκή ε, Ομοσπονδία για τη συνταξιωτική κάλυψη θέλει μια τέτοια προσέγγιση. Όπως ανέφερε ο συνάδελφος, τα εμπόδια είναι η φορολογία και οι κανόνες, οι ρυθμίσεις και υποπτία, οι κανόνες φερεγγιότητας ε, ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Αυτά είναι τα βασικά εμπόδια για να υπάρξει μια ολοκλήρωση και μια προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα. Να σας δώσω άλλο ένα εμπόδιο στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, είναι το πολιτικό εμπόδιο. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, έχουμε κοινή εμπειρία. Υπάρχουν διαφορετικά συναισθήματα στα δεξιά κόμματα και στα αριστερά κόμματα όσον αφορά την προσέγγιση για τη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση. Απλούστατα. Για τα δεξιά κόμματα αλλάζει η κατάσταση, πάει μόνο σε ατομικές συντάξεις, επικουρικά συστήματα κλπ. κλπ. Αριστερά κόμματα. Χρειάζεται συνταξιδότηση σχετική, DB κλπ. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε κατά πόσο χρειάζεται να έχουμε ένα βασικό στεξιδρικό σύστημα. Εμείς πιστεύουμε ότι ναι πρέπει να το έχουμε αυτό. Κοινωνικός στόχος είναι βιώσιμα συνταξιωτικά ταμεία. Και το DC δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε βιώσιμη σύνταξη για όλους στην Ευρώπη. Πρέπει να τεθούν ευρωπαϊκοί στόχοι. Το DB ανεξάρτητα από χρηματοδοτείται. Στη χώρα μας είναι από το δημόσιο τομέα. DB είναι ο στόχος. Αμερική, Βρετανία πάνε από DB σε DC. Γιατί θέλουν υποτική προσέγγιση. Θέλουν τον καλύτερο φορέα. Τον ιδιωτικό φορέα. Είναι οι μέτοχοι Ισχυρή μέτοχοι που συμμετέχουν στα σχήματα. Και είναι πιο ισχυρή που μας πρόχνουν να πάμε από την σε Άρα ίσως να είναι και μια ευκαιρία για την Ευρώπη να αλλάξει. Σας ευχαριστώ. Να διαβάσω τον κατάλογο των ομιλητών που έχουν ζητήσει το λόγο. Όλοι Σμιτ. Dann Herrn Zille, dann äh, Huang Ngox, äh, Frau Thompson, Und zum Schluss Και αν θέλει κανείς άλλο το λόγο. μου λένε ότι και ο κύριος ε, Γκόγκς ε, πρέπει να φύγει σε λίγο, γιατί θα δώσω καθήν το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Euh, ma question s'adresse à Κοιτάξτε. Des Και οι προβλέψεις που γίνονται γίνονται επί δημογραφικής για τα ενεργά μέλη τη κοινωνία σε σχέση με αυτού που ενεργάζονται. Τώρα σαν οικονομολόγος να το δω, υπάρχουν περιορισμοί οικονομικοί, κατακεφαλοποίηση και κατανομή για τη χρηματοδότηση και εξαρτώνται αυτά πολλέ παραμέτρους. Δημογραφικό παράγοντα, το επίπεδο γονιμότητας, μετανάστευσης, παράγοντες που είναι δύσκολο να προβλέψουμε στον ορίζοντα 2050. Οι προβολές όμως εξαρτώνται και από την παραγωγικότητα κάθε ενεργούς μέλους, κάθε εργαζομένου. Και οδηγεί στο δυναμικό, η δραστηριότητα οδηγεί στη δυναμικότητα ανάπτυξης της οικονομίας. Σήμερα είναι αρνητική. Αν η στρατηγική του 2020 Ευρωπαϊκή Ενώσεως πετύχει, θα είχαμε τότε ε, πολύ ψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης από το 1% του 2050. Αν πετύχει τους στόχους, σίγουρα θα έχουμε με την οικονομία της γνώσης 3-4% το χρόνο ανάπτυξη. Τελευταία παράμετρος όσον αφορά τα κατανεμμένα συστήματα είναι το τμήμα του μισθού, το μερίδιο του μισθού, βάσει του οποίου ε, γίνονται, εισπράττονται εισφορές. Και μειώθηκαν οι μισθοί σε όλες τις χώρες του ΩΣΑ και το 2050 η αξία των μισθών δεν ξέρουμε αν θα αποκατασταθεί ή όχι. Ή αν θα ανέβει 1-2% στο 1,2% η αύξηση του ΑΕΠ. Ο ΣΑΤΑ έλαβε αυτά υπόψη Στι προβολές. Διότι δεν νομίζω ότι συμπεριλαμβάνονται. Εν τη αυτή περιπτώσει. οι διάφοροι τρόποι χρηματοδοτήσεως των ε, συστημάτων διευκολύνονται Το άλλο σύστημα, όχι της αντίθε... ε, άντεξε καλύτερα την κρίση. Και οικονομικά και κατάφεραν να αποσβέσουν τα αποτελέσματα της κρίσης. Τα αναγνωρίζουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στην Ευρώπη. Και είναι η βάση των συστημάτων των συνταξιδοτικών στις χώρες του Eurogroup. Ο κ. Σάμεκ το υπενθύμησε. Στον ΩΣΑ ή αλλού υπάρχει ανάλυση όσον αφορά τη διεύρυνση της βάσης χρηματοδότησης του συστήματος του αναλογικού. Πέρα από τη βάση του μισθού, να λάβει υπόψη το οικονομικό εισόδημα για τη χρηματοδότηση αυτού του συστήματος. Um, Κοιτάξτε. Θα Είμαι σύντομος για να απαντήσω σε ένα στοιχείο. Δεν κάνουμε στον ΩΣΑ τέτοιες μακροπρόθεσμες προβλέψεις για δαπάνες σε σχέση με την ηλικία. Αυτό το αφήσαμε στην ομάδα που ασχολείται ε, με θέματα γύρανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δικές τους προβλέψεις κατέτεξαν ότι η γύρανση θα επιδράσει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της επόμενης δεκαετίας και γι' αυτό λοιπόν έγιναν προβλέψεις μέχρι το 2060. Το θέμα με την γύρανση των κεφαλαγορών είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον και υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες κοιτάνε ακριβώς τη σχέση της γύρανσης σε ό,τι αφορά την απόδοση των επενδύσεων. Οι μελέτες που εμπιστεύομαι υποδεικνύουν και καταδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρχει μικρός αρνητικός αντίκτυπος και ότι Πρέπει να σας πω ότι δεν αποδέχομαι τις πιο εφάνταστες ε, προβλέψεις που μιλάνε για ε, τελείως κατάρρευση των ε, συστημάτων και ότι οι επενδυτέ θα πρέπει να πληρώνουν τα συνταξιδετικά του συστήματα, τα συνταξιδετικά του προγράμματα τελείω. Δεν θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ένα ρεαλιστικό σενάριο για το μέλλον. Είναι δύσκολο να προσθέσω κάτι γιατί είμαι πεπισμένος ότι η καλύτερη λύση είναι ένα περίπλοκο σύστημα από, τρίο, από τρεις πυλώνες. Κάναμε τρεις απόπειρες στην Τσεχία να εισάγουμε επαγγελματικά συστήματα συνταξιοδότησης. Τρεις, τρία νομοσχέδια, τα οποία απορρίφθηκαν στο Κοινοβούλιο για ιδεολογικούς λόγους. Υπάρχουν κάποια λογικά επιχειρήματα για κάποιες μεταρρυθμίσεις, αλλά από πλευρά συνδικάτων θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να δώσουμε στον κόσμο την ευκαιρία να είναι ελεύθερος σε ό,τι αφορά το συμπλήρωμα της δημόσιας συνταξής τους, γιατί είναι σαφές ότι τα δημόσια συστήματα θα είναι πιο φτωχά ως προς τον βαθμό αντικατάστασης. Και είναι σαφές ότι στο μέλλον θα είναι δύσκολο να προβλέψουμε αν το 2050 θα δουλεύει ο καθένας μας τρεις ή τέσσερις ημέρες, γιατί σήμερα δουλεύουμε ιστορικά έξι ημέρες. Ίσως να είναι πιο υψηλή η παραγωγικότητα στην κοινωνία και να δουλεύουμε μόνο τρεις-τέσσερις ημέρες. Το ελπίζω. Ελπίζω να υπάρχει τέτοια δυνατότητα ανακατανομή ε, χρημάτων μεταξύ του ενεργού και μη ενεργού πληθυσμού. Ίσως με διαφορετικό τρόπο από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Ίσως λοιπόν να είναι απαραίτητο όχι μόνο να υπάρχουν ε, εισφορές από τις ηλικίες ομάδες, αλλά από τους ε, φόρους. Uh, uh, Πολύ σύντομα. Το ερώτημα νομίζω απαντήθηκε το άλλως. Μια προσθήκη απλώς όσα υπόθηκαν και στην παρουσίασή μου ανέφερα την αυξανόμενη παραγωγικότητα που θα είναι σημαντικό παράγοντα επειδή ο εργαζόμενο πληθυσμό θα συρρυκνωθεί. Και αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό Ιδίω στι χώρε τη Κεντρικής Ευρώπης, να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα στις χώρες μας, τι περισσότερες χώρες μας, το σύστημα έρευνας έχει καταρρεύσει. Δεν γίνονται επενδύσεις για να βοηθηθούν τα ερευνητικά ιδρύματα. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση από τον δημόσιο προπολογισμό. Χρειάζονται επενδύσει, γιατί πολλοί από του επιστήμονε μα έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Θα πάρει χρόνια λοιπόν οι κυβερνήσει να ανοικοδομήσουν το ερευνητικό σύστημα και να φτάσουμε σε ψηλά επίπεδα εάν θέλουμε παραγωγικότητα να αυξηθεί σε κάθε τομέα. Πάντω, οποιοδήποτε κυβερνητικό μέτρο θα εξυπηρετούσε αυτή τη διαδικασία θα ήταν πρόσδεκτο. Κάποια άλλα θα έρθουν ε, με φυσικό τρόπο μέσα από τις ξένες επενδύσεις, κάποια βραχυπρόθεσμα. Πάντως, συμφωνώ ότι αυτή θα πρέπει να είναι από τι πρώτε προτεραιότητε για τη μακροχρόνια στρατηγική μα. Να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των συνταξιδοτικών συστημάτων. Η κυρία Τόμσον και ο Όλη Σμιτ θα σα απευθύνω, θα σας παρακαλέσω να απευθύνετε τι ερωτήσει σα σε ένα μόνο πανελίστα, γιατί δεν θα μα φτάσει ο χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και το πάνελ για τι παρουσιάσει του σήμερα. Είχαμε και ένα άλλο πάνελ για τις διαφορές μεταξύ των γενεών και τώρα μας μιλήσατε και εσείς για τις διαφορές μεταξύ των νέων και των παλαιών κρατών μελών. Εγώ μόλις έρχομαι από μία ακρόαση στην Επιτροπή για την ισότητα των ε, δικαιωμάτων των δύο φύλων σε ό,τι αφορά το δικό χάρτη για τα φύλλα στην Ένωση. Θα ήθελα να υπάρχουν και στατιστικά στοιχεία αναφύλλω γιατί όταν μιλάτε για τις ε, εισφορές ε, σε ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης, ε, μιλάμε για γυναίκες ή για άντρες. Γιατί βλέπουμε ότι η θέση των γυναικών σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις είναι ακόμα χειρότερη. Στη χώρα μου, στη Δανία, οι γυναίκες κατά μέσο όρο λαμβάνουν το 50% των συντάξεων των αντρών. Είμαστε 53% οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αυξηθεί το ποσοστό αυτό όμως. Το 2025 το 10% του πληθυσμού θα είναι 85 ετών και το 90% του πληθυσμού που θα είναι 85 και πλέον ε, ετών θα είναι γυναίκες. Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν το πρόβλημα αυτό. Όλοι Σμιτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από 15 χρόνια όταν ήμουν ε, βουλευτή στην Σουηδία σε μία άλλη ε, σκανδιναβική χώρα, αλλάξαμε τελείως ε, το συμβενταξιωτικό σύστημα από ένα σύστημα παγιασγικό σε ένα σύστημα πιο... Α, ε, σύστημα premium. Και όπως αναφέρατε νομίζω στα έγγραφα του ΩΣΑ, η αυτόματη προσαρμογή των παροχών. Να σας ρωτήσω λοιπόν, επικρίνεται τα συστήματα αυτά, όπου υπάρχει σύνδεση μεταξύ των συντάξεων και της συνολικής οικονομίας, όταν ο μέσος όρος δηλαδή ε, των μισθών μειώνεται, αυτό επηρεάζει και τις ε, συντάξεις. Βλέπω ότι αναφέρατε ότι δεν πιστεύατε ότι θα συμβεί αυτό στη Σουηδία. Συνέβη όμως και φυσικά έχει προκαλέσει ε, μεγάλη αντίδραση. Ποιο άλλο σύστημα λοιπόν υπάρχει, αν, δεν, θεωρείτε ότι δεν είναι καλό το σύστημα αυτό, ποιο άλλο σύστημα υπάρχει, θεωρείτε ότι θα υπάρχουν πιο υψηλή φορολογία, λιγότερη ευημερία, γιατί φυσικά αυτή είναι η μοναδική άλλη εναλλακτική λύση. Πείτε μας λοιπόν, για ποιον είναι η ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος, για τον ΩΣΑ, για τον κύριο Whitehouse. Γιατί από ό,τι βλέπω ασκεί κριτική ο ΩΣΑ αυτό το συνταξιβετικό σύστημα όπου υπάρχουν τέτοιες ε, προσαρμογές και μου προκαλεί έκπληξη αυτό για να απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις. Κοιτάξτε, έχω στον υπολογιστή μου τα στοιχεία και όχι εδώ. Μπορώ να ξεχωρίσω τα εισοδήματα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έχουν ξεκινήσει τρία έγγραφα. Έχουμε τρία έγγραφα. Το ένα εξετάζει τα δικαιώματα εξωτικά για τι γυναίκε που προσέχουν, είναι εκτό αγορά εργασία και έχουν παιδιά. Για άλλα, για ε, συντάξει ενό επιβιώσαντο από το ζευγάρι, αν είναι μια χείρα 85 ετών που έχει μεγάλη διάρκεια ζωή μπροστά τη. Και θα εκπονήσουμε σχετικά έκθεση το μέσα του 2011 όταν τελειώσει η δουλειά, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες και έχει προτεραιότητα στα συγκεκριμένα ερωτήματα για τη Σουηδία. Δεν επικρίναμε τους μηχανισμούς. Εγώ είπα ότι χρειαζόταν μια νέα ανάλυση, κυρίως λόγω των πολιτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται στη Σουηδία και στη Γερμανία όπου είναι παρόμοιες προσαρμογές για τη βιωσιμότητα που γίνονται στα δεξιωτικά συστήματα. Ένα συγκεκριμένο θέμα στη Σουηδία και το εξή. Ένα τρόπο προσμέτρηση φερικιότητα του συστήματο συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία ενεργητικού, την αξία των στοιχείων ενεργητικού του ταμείου. Περίπου ένα τρίτο των στοιχείων παθητικού το ίδιο, η ίδια ανάλυση γίνεται και στη Φιλανδία που εκεί γίνεται μερική χρηματοδότηση. Αν συγκρίνουμε αυτά που έγινε στον Καναδά με αυτά που έγινε στη Σουηδία, έχει παρόμοιο μηχανισμό ο Καναδά. Εκεί έχει την απόσβεση του κόστου τη κρίση, των συνεπειών τη κρίση, <clears throat> επί τη αξία του ταμείου πάνω στον ανορίζοντα πεντηκονταετή. Ενώ οι κανόνε στη Σουηδία είναι συγκεκριμένοι, ότι η αξία τη αγορά μπαίνει στην εξίσωση και τα ευεργετήματα πρέπει να μειωθούν τον επόμενο χρόνο δεν επικρίνουμε τους μηχανισμούς. Λέμε ότι αντιμετωπίσαμε μια κρίση και δεν λειτουργήσαν οι μηχανισμοί. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι κανόνες δεν τηρήθηκαν στη Σουηδία, η μείωση κατανεμήθηκε σε μια χρονική περίοδο όπως και στη Γερμανία. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται νέα ανάλυση, διότι η πρώτη φορά που έπληξε η κρίση ο αυτόματος χαρακτήρας τους δεν λειτουργήσε τελικά. Thank Κύριε Γκίγκολτ, ευχαριστώ Να πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι δεν έγινε δελεχής ανάλυση των συνεπειών της κρίσεως επί των συνταξιδοτικών συστημάτων κυρίως από εκείνον που περίμενα να το κάνει, τον εμπειρογνώμονα του ΩΣΑ. Κατά την άποψή μου, φτάσαμε στο σημείο τήξης του συστήματος, των νομισματικών συστημάτων των κεφαλαίων Θα πρέπει να συναγάγουμε συμπεράσματα. Λόγω παρεμβάσεων των κυβερνήσεων, απεφεύχθη το χειρότερο. Τι σημαίνει αυτή η εμπειρία μας από την κρίση. Τι συνεισφορά θα έχει στην αναδιάθρωση των συνταξιωτικών συστημάτων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούσατε. Οι προβολές. Τα στοιχεία που έδειχαν πως μειώθηκαν τα ποσοστά κερδών των ταμείων. Είναι παλαιού τύπου προσέγγιση που δεν λαμβάνει υπόψη του συστημικού κίνδυνου. Ο συστημικός κίνδυνο είναι δυσκολότερο να ποσοτικοποιηθεί. Αυτό που θα ήθελα να δω θα ήταν πιο συστηματική ανάλυση για το πώς θα οικοδομήσουμε τα συνταξιωτικά συστήματα μετά την εμπειρία των μεγάλων κινδύνων μετά την κατάρρευση του χρηματοσυστικού συστήματος άλλη προσέγγιση του κινδύνου από αυτήν που αναλύθηκε όσον αφορά και περιεγράφει όσον αφορά την Ανατολική Ευρώπη. Το ερώτημά μου σχετίζεται με το νέο πολιτικό δίλημα το οποίο δημιουργήθηκε από την κρίση. Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κινήθηκαν, προσπάθησαν να βρουν μια λύση απέναντι σε αυτό το δίλημα. Οι επενδύσεις των συνταξιωτικών ταμείων είναι διαφορετικές στις πλούσιες χώρες και διαφορετικές στις στοχές. Οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση τη χώρα και να επηρεάσει τις δυτικές χώρες. Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία. Αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και ίσως δεν είναι τόσο καλές οι αποφάσεις των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των συνταξιοδοτικών ταμείων. Έχουν γίνει πολλές επενδύσεις από τα σκανδιναβικά κράτη στα συνταξιοδοτικά ταμεία των βαλτικών χωρών και πολύ συχνά τα δάνεια ε, γίνονται σε ευρώ, χορηγούνται σε ευρώ και όχι σε εθνικά νομίσματα. Πρέπει λοιπόν να μειωθούν οι επενδύσεις του δεύτερου πυλώνα για να σωθεί ο πρώτος. Ο πρώτος πυλώνας έχει λιγότερα έσοδα. Αυτό γιατί μειώνονται οι μισθοί. Και πολλοί είναι άνεργοι. και τα νοικοκυριά μας θα πρέπει να αποπληρώσουν τα χρέη τους έναντι των σκανδιναβών επενδυτών και αυτοί οι επενδυτές δεν πρέπει να κάνουν τόσο μεγάλες προσαρμογές βιωσιμότητας που ανέφερε ο κύριος Whitehouse. Ή θα πρέπει να δημιουργήσουμε τα δικά μας συνταξιωτικά συστήματα διαφορετικά. Νομίζω ότι η πρώτη μας συνταξιωτικα συστηματα διαφορετικα Νομίζω ότι η προτεραιότητα απευθύνεται στην και οι και στου δύο. Καταρχά, για. Για το γενικότερο ερώτημα, για τη σχέση τη κρίση με τα συνταξιδοτικά ταμεία, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα συνταξιδοτικά ταμεία γενικώ δεν είχαν τόσα τοξικά περιουσιακά στοιχεία όπως τα χρεόγραφα που είχαν χρησιμοποιηθεί στην υπόλοιπη χρηματοπιστωτική αγορά. Είχαμε περίπου 3% τέτοια στοιχεία στα, στα ταμεία. Τα συνταξιδοτικά ταμεία κυρίως στα κυβερνητικά ομόλογα, στα αξιόγραφα και στα κίνητα επενδύουν. Βέβαια το χρηματιστήριο δεν ήταν εξαιρετικό ούτε πέρυσι, αλλά τα συνταξιδοτικά, τα συνταξιδοτικά ταμεία αποφεύγουν τους συστημικούς κινδύνους. Και ένα από τα βασικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής ήταν ότι όταν ο κίνδυνος τα επιτόκια μάλλον για δευτερουσιακά περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με διαφορετικές τάξεις ε, ε, και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων έδιναν και διαφορετικά κέρδη. Εδώ ο ποσοστό έκπτωσης ήταν ε, Διαφορετικό βεβαίω από κατηγορία σε κατηγορία, γι' αυτό και αν με την κρίση επηρεάστηκε ακόμη περισσότερο, γι' αυτό βεβαίω πολλέ απρόβλεπτε συνέπειε είδαμε. Και σίγουρα η κατάσταση της χρηματοπιστωτικής αγοράς επηρέασε. Maybe one provoke, uh, consider... Να πούμε και να το σκεφτούμε αυτό. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό για τα μελλοντικά σταξιδικά συστήματα. Επειδή ο κόσμος μας ε, πολλαπλασιάζεται, επειδή αυξάνεται, είναι δύσκολο να πετύχουμε το μέσο στο ανάπτυξης. Αν ε, όλος ο κόσμος ε, αξιοποιούσε αυτό το κόστος, αυτή την ανάπτυξη μόνο για τα δυτικά συστήματα. Είναι σαφές ότι είναι το μοναδικό κριτήριο που μπορούμε να ακολουθήσουμε και μπορούμε ίσως αν θέλετε να συζητήσουμε ποια είναι καλύτερα συστήματα τα δημόσια ή τα ιδιωτικά συνταξιωτικά συστήματα. Εγώ θα ήθελα να ανανεωθεί ο ρόλος των δημοσίων συστημάτων DB, γιατί ουσιαστικά αποτελούν τη μοναδική προστασία από τη φτώχεια και αν λάβουμε υπόψη και τις διαφορές μεταξύ των μισθών γυναικών και ανδρών, γίνεται συζήτηση για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά επίσης την κατανομή των συνταξιβετικών ε, δικαιωμάτων, όπως γίνεται στην Ελβετία. Γίνεται κατανομή κάθε χρόνο μεταξύ των ε, συζύγων. δεν υπάρχει μία ενιαία προσέγγιση, ένα ενιαίο σύστημα στην Ευρώπη για, την, για τα συνταξιωτικά συστήματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές και εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα για τις ε, συντάξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει και σχετική ατζέντα. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν να διευκρινίσουμε τι σημαίνει το κοινωνικά δέον εισόδημα και η τελευταία απάντηση από την κυρία Σιωριέλ. Αν δούμε τι γίνεται στο δεύτερο πυλώνα στην περιοχή μας, βλέπουμε ότι και η εκχώρηση των ε, είναι πολύ σαφώς ρυθμισμένες και ποιες, ε, πιο πολλές επενδύσεις γίνονται στο ιστορικό της χώρας σε τοπικό επίπεδο, αλλά και επειδή γενικά τα αξιόγραφα είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο, καλό θα ήταν να αλλάξουμε τα όρια αυτά και να βάλουμε πιο υψηλά πλαφόν. Θεωρώ επίσης ότι θα ήταν καλό όντως να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό θα βοηθούσε και θέματα κινητικότητας που περιορίζεται σήμερα στο ιστορικό της Ευρώπης, αλλά αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα εμπόδιο σε ό,τι αφορά τα συνταξιβετικά συστήματα. Ως προς τον τύπο των προϊόντων που μπορεί να παρέχονται μέσω του DB και του DC, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να επιλέξουμε ένα από τα δύο θεωρώ ότι ο συνδυασμός των δύο θα ήταν πιο σωστός, ιδιαίτερα για το δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας ή για ένα ελάχιστο επίπεδο στους πυλώνες. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε ότι το σύστημα πολλαπλών πυλώνων είναι πολύ διαφορετικό. Για παράδειγμα, το μοντέλο της Παγκόσμιας Τράπεζας με τρεις ή πέντε πυλώνες θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο η Ένωση της Γενέβης έχει τέσσερις πυλώνες. Υπάρχουν διαφορετικές λοιπόν λύσεις και κοιτώντα τις χώρες της Δυτικής, Ευρω... της Δυτικής Ευρώπης βλέπουμε ότι οι πυλώνες έχουν διαφορετικό νόημα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώσαμε την σημερινή μας ακρόαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές μας, τους προσκεκλημένους και του πρώτου πάνελ και του δεύτερου πάνελ. Φυσικά πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά, αλλά όπως είπατε και εσείς θα έχουμε τροφή για σκέψη. Έχουμε λάβει καινούργιε ιδέε, τι οποίε σίγουρα θα αξιοποιήσουμε στι μελλοντικέ μα εργασίε. Σα ευχαριστώ και θα παραμείνουμε σε επαφή. Τη Δευτέρα έχουμε στι 4 το, το απόγευμα την επόμενη συνάντησή μα.